Good afternoon, uh, uh, Καλώς ήλθατε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Παίρναμε και πάλι στο σημείο 9 που είναι οι ανακοινώσεις της Προέδρου κανονικά, αλλά θα γίνει του Προέδρου, γιατί το είχαμε αναβάλει το σημείο αυτό μέχρι απόψε. για τον οικονομικό διάλογο με τη Γαλλία μας πληροφορήσανε ότι για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη συνάντηση με τον, Υπουργό, με τον Πρωθυπουργό κύριο ε, Ολάντ. Ο Υπουργός Οικονομικών κύριος Μοσκοβιτσί θα μπορέσει να έρθει στη συνάντησή μας που προβλέπεται στις 13 Νοεμβρίου για τον διάλογο αυτό. Προβλέπεται τώρα να γίνει μια συνάντηση στις 12 Φεβρουαρίου το απόγευμα του 2014. Η Επιτροπή Εξωτερικών επίσης της ε, Ολλανδικής Νομοσπονδίας, 25 μέλη και το προσωπικό τους, θα έρθουν στις 13 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουν να συναντηθούν με εμά, με την Επιτροπή ΙΜΚΟ, ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσοι ενδιαφέρονται για τις σχέσεις με την Ολλανδία, με την Ελβετία, συγγνώμη, και κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την φορολογία, το τραπεζικό απόρριτο κτλ. προσκαλούνται να συναντήσουν τους Ελβετούς κοινοβουλευτικούς από τις 9 ως τις 10, 13 Νοεμβρίου. Το επαναλαμβάνω. Η γραμματεία μας θα σας στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περαιτέρω πληροφορίες εν καιρό για εν εξελίξη τριλόγους, τριγωνικούς διαλόγους. Ο τελευταίος έγινε 22 Οκτωβρίου τον, στο Στρασβούργο και πρόκειται για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανακεφαλαιοποίηση και την ευκαμψία καθώς και τα εργαλεία για την σταθερότητα στα κρατικά οικονομικά. Επίσης συζητήθηκαν και θέματα εσωτερικά και ο τελευταίος τριγωνικός διάλογος θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου σε σχέση με τον τριγωνικό διάλογο Omnibus. Ο 12 ο τέτοιο διάλογος έγινε στην 5η 24 Οκτωβρίου. Δεν υπήρξε καμία πρόοδος ουσιαστικά για κανένα θέμα. Η 24 οκτωβριου δεν υπηρξε καμια προοδο ουσιαστικα για κανενα θεμα η ομαδα διαπραγματευση του Κοινοβουλίου έκανε πολλά σχόλια σε σχέση με το κείμενο της Προεδρίας σε ό,τι αφορά τι τις εγγύησει. και τα σχόλια αυτά περιλάμβαναν μια αίτηση για περαιτέρω ε, διευκόλυνση της επίτευξης μιας λύσης. Η Κομισιόν ήταν θετική για πολλά από τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά η Προεδρία εξέφρασε τις ανησυχίες της ότι οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να αποσταθεροποιήσει το πακέτο. Και επίσης για το έγγραφο για τα οικονομικά εργαλεία δεν υπήρξε κάποια θετική αντίδραση από την Προεδρία. Ο 13ος διάλογος θα γίνει 13 Νοεμβρίου. Πάμε στο σημείο 14 της ημερησίας διάταξης. Η ακρόαση για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σε χώρες που μαστίζονται από την κρίση είναι τμήμα μια σειρά από δημόσιε ακροάσπων που διοργανώνει η Επιτροπή μας. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτό το... αυτή η συνάντηση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μια επίσημη έρευνα για τα θέματα της κρίσης. Έχουμε ζητήσει την έγκριση να δημιουργήσουμε μια έκθεση πρωτοβουλία σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ελπίζουμε ότι αυτή η ακρόαση μπορεί να βοηθήσει να δώσει στοιχεία για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης από τη στιγμή που θα τύχει έγκρισης. Θέλω να καλωσορίσω ε, ομιλητές μας. Τα βιογραφικά τους σας έχουν αποσταλεί με email και σας υπενθυμίζω ότι ο στόχος της σημερινής ακρόασης να κάνουμε μια επισκόπηση των επιτυχιών και μη επιτυχιών των δράσεων αυτών στις χώρες ε, κρίσης γιατί πολλές φορές αμφισβητούνται οι ενέργειες που έγιναν από την Τρόικα και επίσης και η δημοκρατική νομιμότητα των μέτρων ε, αμφισβητείται. Μας ενδιαφέρει και ο μακροχρόνιος αντίκτυπος στις χώρες αυτές και πώς θα μπορούσαν οι χώρες αυτές να ωφεληθούν από μια διάφανη και ουσιαστική επισκόψη και ανάλυση των μέτρων αυτών και να τονίσουμε ποια μέτρα έχουν λειτουργήσει και σε ποιο πλαίσιο. Έχουμε δύο πάνελ. Το πρώτο <clears throat> θα εξετάσει την, ε, το βρόχο ανάδραση μεταξύ κρατικού χρέους και τραπεζικού τομέα και το δεύτερο θα αντιμετωπίσει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την κοινωνική διάσταση στις χώρες κρίσης. Θα ξεκινήσουμε με μία σύντομη παρουσίαση από τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες μας και θα ακολουθήσει μία διαδικασία Catch the Eye και θα ακολουθήσει και και θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ έχουμε ένα κατάλογο ομιλητών. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως με τον καθηγητή Ζωριόν, ο οποίος είναι καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Ο κύριος Ζωριόν έχει πέντε λεπτά στη διάθεσή του.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 I start? Can I be heard? Ακούτε να ξεκινήσω. Καταρχάς κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι μου είπαν ότι είχα 10 λεπτά στην διάθεσή μου. Όντως έχω 10 λεπτά. Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Έδωσα στην ε, ομιλία μου τον τίτλο «Το μέλλον της Ευρωζώνης από την άποψη των επιτοκίνων». Το μέλλον της Ευρωζώνης ε, μπορεί να προσεγγιστεί σε ένα λογικό πρόβλημα. Εάν δεν επιληθεί, τουλάχιστον μπορεί να διευκρινιστεί όταν εξετάζεται το θέμα από την άποψη του τοκομεριδίου του κρατικού χρέους. Στα πλαίσια της οικονομικής ζώνης, εκεί που υπάρχει ένα νόμισμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα και μόνο το κομερίδιο για κάθε υποχρεωτική λήξη. Οι ιδρυτές πατέρες της Ευρωζώνης υπέθεσαν ότι κάτι τέτοιο θα συμβαίνει και για τη ζώνη. Τουλάχιστον μακροπρόθεσμα θα συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν πρόβλεψαν ότι ο κίνδυνος διακοπής πληρωμών θα φορούσε κάποιο μεμονωμένο μέλος της περιοχής, ούτε θα μπορούσε να θεωρηθεί μια εναλλακτική λύση επιστροφής στο παλινό νόμισμα. Το γεγονός ότι ότι τα τοκομερίδια αλλάζουν σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται στην Ευρωζώνη είναι ένα ε, σύμπτωμα των προβλημάτων. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τοκομεριδίου κρατικού χρέους. Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τρία στοιχεία που αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τις οικονομικές αλλά και τις πολιτικές ε, συνθήκες των μεμονωμένων χωρών στη ζώνη ε, ρευστότητα, επιστοτικό πριν και πριν μετατρεψιμότητα. Όταν θα αναφερθώ στο τοκομενίδιο που έχει σχέση με το κρατικό χρέο μια ειδική, ιδιαίτερη ημερομηνία λήξη, αναφερθώ σε ένα επιτόκιο που αποτελείται από τα τρία αυτά στοιχεία, μολονότι το πιστοτικό πρίμε και το πρίμε μετατρεψιμότητα ε, έχουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μηδέν αξία. Το πριν ρευστότητα αποτελεί το μέρο του επιτοκίου που δεκτοροπίζει το γεγονό ότι ένα εργαλείο χρέου ε, δεν είναι χρήματα, αλλά ένα ε, βασικό αγαθό το οποίο θα μετατραπεί σε χρήματα. Είναι η τιμή η οποία εκφράζεται ως ε, επιτόκιο για κάτι τέτοιο. Το πριν ρευστότητα για μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξη ενό νομίσματο καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ των υποψήφιων δανειστών και των υποψήφιων ε, δανειζόμενων. Η προσφορά και η ζήτηση, η ζήτηση αποτελεί ένα από αυτού του παράγοντε από τη στιγμή που αυξάνει τον ανταγωνισμό είτε μεταξύ δυνητικών δανειστών δανειζόμενων ε, ή μεταξύ δυνητικών δανειστών. Το πριν ρευστότητα διαφέρει μεταξύ των νομισμάτων και αυτό αντικατοπτρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομική ζώνη. Αυτές οι διαφορές ε, ανοίγουν ευκαιρίες διευθυνσίας ενός συγκεκριμένου τύπου που ονομάζεται carry trade, arbitrage επιτοκίων. Ε, μπορούν να, ο δανεισμός μπορεί να γίνει σε ε, ένα συγκεκριμένο νόμισμα. Το, πρίμα, το πιστοτικό πρίμα ζητείται από τον δανειστή σε μια διασφάλιση, σε ένα πρίμα διασφάλιση σε σχέση με το κίνδυνο που υπάρχει για διακοπή πληρωμών. Αυτά θεωρούνται ε, πιστοτικά συμβάντα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αγορά για τα πιστοτικά πρίμα. Τα swaps, τα CDS, η αγορά των CDS, αλλά και τα ακάλυπτα τα CDS. Το πριν μετατρεψιμότητα ε, καλύπτει το κίνδυνο τα χρήματα που υπάρχουν σε ένα νόμισμα θα επιστραφούν σε ένα διαφορετικό νόμισμα. Ε, για παράδειγμα, μετά από μια επιστροφή στη δραχμή, στο τα κτλ. Στο σκούδο κτλ. Θα ε, επιστρέψω τώρα στην Ευρωζώνη. Το κομερίδιο κρατικού χρέους στην Ευρωζώνη, εάν η Ευρωζώνη είναι η πιο οικία περίπτωση όπου το, το κρατικό χρέος ε, ε, ε, ενός νομίσματος συνδυάζεται με πάνω από ένα το κομερίδιο, η αρχή παραμένει ότι το κρατικό χρέος σε ένα ε, ε, σε μία λήξη ε, προθεσμίας αφορά ένα πριμ ρευτότητας. Μέσα στην Ευρωζώνη το πριμ ρευτότητας για μία συγκεκριμένη λήξη, ε, ημερομηνία λήξης θα μπορούσε να υπολογιστεί εξετάζοντας τα επισόγια. Και οι αγορές θεωρούν ότι είναι μηδενικός ο κίνδυνος στη Γερμανία να υπάρξει τάση πληρωμών. Ε, κατά τον ίδιο τρόπο, οι κεφαλαιογικέ αγορέ θεωρούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να εκφράσει επιθυμία να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Ε, δεν θεωρείται κάτι ε, πιθανό. Συνεπώ, δεν υπάρχει πρίμε μετατρεψιμότητα που να έχει σχέση με το κρατικό χρέο τη Γερμανία. Σε ένα άρθρο με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2012 στο New York Review of Books με τίτλο The Tragedy of the European Union and How to Resolve It, ο, ο ε, ε, αναφέρει ότι η Γερμανία θα πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο, τα τοκομερίδια της ε, Γερμανίας ε, θα αρχίσουν να συμπεριλαμβάνουν ένα πρίμε Σε Αυτό θα έχει αρνητική αξία και θα μειώσει το επιτόκιο του όλου το κομεριδίου από τη στιγμή του ευρώ της Ευρωζώνης χωρίς τη Γερμανία θα υποτιμηθεί. Από τη στιγμή που τα τοκουμερίδια του γερμανικού κρατικού χρέους θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σημείο αναφοράς ε, σε ό,τι αφορά το πριν ρευστότητα, ε, το αποκαλούμενο spread του τοκομερεδίου για ένα άλλο κρατικό χρέος είναι το άθροισμα, το, πριμ, ε, το πιστοτικό πριμ και το πριμ μετατρεψιμότητας. Μόλις ε, Άρχισε να γίνεται πιστευτό κάτι τέτοιο και τη απουσία οποιαδήποτε δέσμευση ότι αυτή η χώρα δεν θα εγκαταλείψει την ζώνη, το η τιμή ε, των ε, πριν αυξήθηκε πάνω από το 0. Μία κέντρο, φυγόκεντρος ε, δυναμική ξεκίνησε για αυτή τη χώρα και συνεπώς έπαψε πλέον να υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Η έλλειψη εμπιστοσύνη στην ικανότητα μιας χώρας να σταθεί στο ύψος των οικονομικών υποχρεώσεων αυξάνει την τιμή της, του, πριμ, του πιστοτικού πριν. Ε, αμφιβολίες ε, που αφορούν ε, την αξιοπιστία οδηγούν στο να υπάρχουν περαιτέρω αμφιβολίες. Η τιμή του πριμ μετατρεψιμότητας προστίθεται σε αυτό του, στο πιστοτικού πρίμα ε, στα πλαίσια του τοκοπεριδίου που απαιτείται από τις κεφαλαιουχικές αγορές για δάνεια. Θα αναφερθώ τώρα στην, ε, στο καταστροφικό δίκτυ ε, ε, κρατικού χρέους και τραπεζών. Μία αρνητική επίπτωση έχει σχέση με τη λογική των πριν πιστώσεων και μετατρεψιμότητας. Ε, αναφέρομαι σε ένα άρθρο με τίτλο The Disaster Sovereign Banking Nexus, όπου, βάσει του οποίου οι εμπορικές τράπεζες θα ε, στηρίξουν το κρατικό χρέος των ε, τραπεζών. Ο λόγος είναι εύκολα κατανοητός ακόμα κι αν φαίνεται κάτι το παράδοξο. Για μια κόρια τράπεζα και τα δύο ε, πρίμε του κρατικού χρέους ε, μεταφράζονται απλά και μόνο σε περιθώρια κέρδους. Το πιστοτικό πρίμα, ε, εάν κηρύξει στάση πληρωμών μια χώρα, οι εμπορικέ τράπεζες είναι πιθανόν να γίνουν αφαιρέγγιες, αλλά θα διασωθούν είτε μέσω της διαδικασίας του bail-in ή του bail-out. Με, πριν εάν επανέλθει μία χώρα στο παλιό νόμισμα, οι εμπορικέ τράπεζε θα κάνουν ακριβώ το ίδιο. Το πριν μετατρεψιμότητα δεν θα μπορεί πλέον να εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Και θα, ε, ε, το αποτέλεσμα θα είναι κέρδο. Ε, ε ε, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με άλλους τύπους έκθεση που περιορίζονται στις τράπεζες το 25% του επιλέξιμου κεφαλαίου, οι τράπεζες μπορούν να αγοράζουν κρατικό χρέος ε, σε όποια ε, ύψος θέλουν. Δεύτερος, όταν αγοράζεται το κρατικό χρέος οι τράπεζες δεν θα πρέπει να βάλουν κατά μέρος μετοχικό κεφάλαιο. Επειδή μια κεντρική τράπεζα είναι ο τελικός δανειστής για τις εμπορικές τράπεζες μιας χώρας, υπάρχει de facto με ένα κοινό πεπρωμένο σε ό,τι αφορά μια κεντρική τράπεζα τράπεζα και τις εγχώριες τράπεζες με τις εμπορικές τράπεζες που συσσωρεύουν όλο και μεγαλύτερες, ε, περισσότερο ε, κρατικό χρέος, εκτίθενται σε ε, μία υποτίμηση. Κάτι τέτοιο δημιουργεί μία σπήρα προς τα κάτω. Υπάρχει αρνητική επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο των εμπορικών τραπεζών και το φάσμα της αφαιρεγγιότητας αυξάνεται ενώ το, το γεγονός ότι πρόκειται για μια μη υγιή κατάσταση αυξάνει, αυξάνει το πιστοτικό κίνδυνο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Σας παρακαλώ διαβάστε πιο αργά γιατί οι διερμηνείς έχουν πρόβλημα να σας παρακολουθήσουν. Ο λέει ο ότι οι διερμηνείς έχουν ένα αντίγραφο της ομιλίας του παρόλα αυτά το εκτιμούσαν πάρα πολύ αν διάβαζε λίγο πιο αργά. να καταλήξω στο συμπέρασμά μου που αφορά τις επιλογές της Ευρωζώνης σε μια σειρά από συμβάντα που ξεκίνησαν τον, τον χειμώνα του 2009 η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και μετά η Ισπανία και η Ιταλία επλήγησαν η μία πίσω από την άλλη σε ένα τέτοιο βαθμό που το κρατικό χρέος των τρίτων πρώτων χρονών χρειάζεται, χρειάστηκε να ε, από την έκδοση στις κεφαλουχικές αγορές από τη στιγμή που τα, πριν, τα ψωτικά πριν και τα πριν μετατρεπτιμότητα έφτασαν τέτοια επίπεδα που οι χώρε δεν ήταν πλέον σε θέση να αποπληρώσουν το τοκομερίδιο που απαιτούσε η αγορά. Η κοινότητα των χωρών ε, που γλίτωσαν, ε, διασώθηκαν στην ε, Ευρωζώνη, ανέλαβαν με τη βοήθεια του Διεθνού Ζωμεζατικού Ταμείου. Η Ιρλανδία λέει ότι θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στι κεφαλαιοχικέ αγορέ το Δεκέμβριο του 2013. Μόνο η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα απαιτήσουν περαιτέρω περαιτέρω ε, υποστήριξη, ενώ η Κύπρος βρίσκεται σε μια, είναι μια οριακή περίπτωση. Το ερώτημα που παραμένει αφορά τις φερεγγιότητες Ευρωζώνης στο σύνολό της. Με την ενδεχόμενη εμφάνιση περαιτέρω τυχημάτων μέσα στη ζώνη, ε, η οποία έχει πληγεί από το 2009, παραμένει το ερώτημα για το προβλέψιμο μέλλον ω προ την ικανότητα των φερέγγιων χωρών ε, μέσα στη ζώνη να υποστηρίξουν σε μια κοινή προσπάθεια τι χώρε εκείνε που έχουν χάσει την πρόσβαση στι κεφαλαιοχικέ αγορέ λόγω τη υπερβολική αύξηση του, πριμ, του πιστοτικού πριμ και του πριμ μετατρεψιμότητα που ζητήθηκε από τι κεφαλαιοχικέ αγορέ. Το γενικό ερώτημα τη Ευρωζώνη στην ουσία στι μέρε μα είναι για το κατά πόσον η αλληλεγγύη που επιδεικνύεται από φερέγγιε χώρε ε, ε, εξασφαλίζει τη φερεγγιότητα της ζώνης στο σύνολό της. πρώτη περίπτωση, ε, η πρώτη περίπτωση είναι και πιο θετική, ότι η γενική φερεγγιότητα της Ευρωζώνης ε, σε αυτή την περίπτωση το δημοσιονομικό πλαίσιο θα παραμείνει, το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο θα παραμείνει υγιές από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει αύξηση στα δύο, στα δύο πριν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επαναεπιτευθεί η ισορροπία όλης της Ευρωζώνης στο φως των νέων περιστάσεων. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή που είναι η πιο θετική που θα μπορούσε να προβλεφθεί για την Ευρωζώνη, παραμένουν στην ουσία σταθείς οι συνθήκες και πάρα πολύ ευμετάβλητες. Η δεύτερη περίπτωση είναι η αρνητική. Στην περίπτωση αυτή η Ευρωζώνη στο σύνολό της θα μπορούσε να είναι αφαιρέγγια. Παρόλε τι κοινέ προσπάθειε, οι φερέγγιε χώρε έχασαν την δυνατότητα που είχαν να παράσχουν εγγυήσει στις προβληματικέ ε, χώρες χωρίς αυτόματα να διακυβεύσουν τη δική του φρεγιότητα. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική Λύση είναι παρακάτω. Να δημιουργηθεί μια μειωμένη περιοχή γενική αφαιρεγγιότητα μετά από την αποχώρηση των αφαιρέγγιων εθνών ε, και ε, οι οποίε θα καταφύγουν ε, στην, διακοπή των πληρωμών και αναδιάρθρωση του κρατηγού χρέου και επιστροφή στο παλιό νόμισμα το οποίο θα υποτιμηθεί σε σχέση με το ευρώ και θα επιτρέψει μια, ένα ξεκίνημα από το μηδέν. Το δεύτερο είναι να προγραμματιστεί μια γενική ε, ε, διακοπή πληρωμών στην Ευρωζώνη, μια αναδιάρθρωση του χρέου στο σύνολό του και μια κοινή προσπάθεια μέσω μιας κοινή αντιμετώπιση μέσα στη ζώνη. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσα στα πλαίσια μιας φεντεραλιστική ε, ε, ομοσπονδιακή αντιμετώπιση. Αυτή η δεύτερη προσέγγιση επιλύει διαπαντό την εγγενή αστάθεια και μεταβλητότητα της Ευρωζώνης υπό την παρούσα συνθήκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγήτα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κωσέφιο Παντεθέο. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να είμαι δυσάρεστος. Θα ήθελα να υπενθυμίσετε στους ομιλητές ότι δεν βρισκόμαστε σε επιστημονικό συνέδριο εμπειρογνωμόνων. Είμαστε εκλεγμένοι βουλευτές, προσπαθούμε να καταλάβουμε να βοηθηθούμε από αυτά που μπορούν να μας πούν οι εμπειρογνώμονες. Δεν έχει κανένα παιδαγωγικό αποτελέσμα να έχει ε, ένας ε, ομιλητής ένα λόγο που τον διαβάζει με μεγάλη ταχύτητα που λαχανιάζουν οι διερμηνείς για να προλάβουν να πούνε κάτι ακόμα και έχουν το κείμενο στα χέρια τους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει να πάρουμε κάποιο μήνυμα από τους ομιλητές. Και νομίζω ότι ο χρόνος που χρησιμοποιούν οι ομιλητές θα πρέπει να μεταφέρει μηνύματα και όχι να μας διαβάζει ατέρμονα κείμενα για 10 λεπτά ένα κείμενο από το οποίο εγώ δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα και πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γοζές. Κύριε Λάγκε. Νομίζω ότι ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Γκοζές. Πράγματι δεν μας προσφέρει πάρα πολύ σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης όταν ακούμε για θεωρητικά σενάρια. Το, τα σενάρια του κυρίου Γεωριών για μένα είναι και τα δύο μη ρεαλιστικά. Η Ευρωζώνη είναι ένα βαθιά πολιτικό εγχείρημα και δεν έχει νόημα να μιλάμε για εναλλακτικά σενάρια. Ούτε το σενάριο 1 που λέει ότι το μεγαλύτερο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα φύγει από την Ευρωζώνη, ούτε βέβαια το δεύτερο που λέει ότι η Ευρωζώνη θα διαλυθεί τελείω στα εξών συνετέθη. Δεν είναι αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει σήμερα. Εμεί θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ και θέλουμε να δούμε κάτω από ποιε προποθέσει είναι δυνατόν τα κράτη τα οποία έχουν αντιμετωπίσει θέματα υπερχρέωσης θα μπορέσουν να ξαναβρούν την ευρωστία τους και την αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών. Είπε ο καθηγητής Γιώριον ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει σωστή διαχείριση του χρέους. Είναι απαραίτητο τα... να εξασφαλίσουμε κάποια ισορροπία σε αυτά τα οποία δίδονται και σε αυτά παίρνονται από τις χώρες αυτές. Τι θα ήθελε να πει ο κύριος Γιώργιον για την υπερχρέωση της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μας βοηθάνε τέτοιου είδους ε, εναλλακτικά σενάρια και δεν είναι χρήσιμα για μας. Ευχαριστώ κύριε Λάγκε. Ο κύριος Κοζές ζήτησε το λόγο για ένα διαδικαστικό θέμα. Εσείς μπορείτε να λάβετε το λόγο στη συνέχεια στη συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Γιώργιον να λάβει υπόψη τα σχόλια του κυρίου Λάγκε και θα επανέλθουμε στην, στο τέλος της συζήτησης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντεθ από την ε, Σχολή Επιχειρήσεων ΙΕ της Μαδρίτης. Σας παρακαλώ να παραμείνετε σε τα 10 λεπτά και ή δυνατόν να είσαστε προσεκτικός με την ταχύτητα της ομιλίας σου γιατί θα πρέπει η διερμηνία να μπορέσει να σας παρακολουθήσει. Microphone. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην μιλάω γρήγορα και να μιλάω αρκετά δυνατά για να με ακούσουν όλοι. Καταρχάς, ε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ε, δεν θα πω ε, ευγενικά λόγια ευχαριστειών, θα πάω κατευθείαν στο θέμα που μας απασχολεί. Έχω κάποιο πρόβλημα με τον τίτλο της ακρόασης «Επιτυχίες και αποτυχίες στις χώρες που βιώνουν κρίση». Ο τίτλος αυτός αγνοεί το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Όχι διότι δεν υπάρχει κρίση σε κάποιες χώρες, αλλά διότι ε, ο σχεδιασμός της Οικονομικής και Νομισματικής ε, Ένωσης είναι εσφαλμένος. Έτσι όπως έχει σχεδιαστεί αυτή η ΟΝΕ αυτή τη στιγμή δεν θα είναι βιώσιμη όσο ε, και αν συμφωνούν οι αγορές για το τι θα γίνει βραχυπρόθεσμα. Θα ήθελα λοιπόν εν συντομία να σας ε, εφιστήσω την προσοχή στα βασικά προβλήματα που υπάρχουν κατά τη γνώμη μου. Έχουμε λοιπόν καταρχάς ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, την οποία καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της οποίας η ανταπόκριση και η αντίδραση στην κρίση έχει γίνει αντικείμενο πολύ μεγάλων επικρίσεων. Το θέμα όμως είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει ασφαλές στοιχείο ενεργητικού ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορεί να υπάρξει νομισματική πολιτική. Αντίθετα με ό,τι ε, συμβαίνει σε άλλα μέρη του πλανήτη μας. Ε, τα στοιχεία ενεργητικού ε, μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πολλούνται και αγοράζονται και δεν έχει την πολυτέλεια αυτή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να παρεύει μέσω κρατικών ομολόγων εθνικών και ε, δεν έχει στοιχεία ενεργητικού για να διεξάγει νομισματική πολιτική στην Ευρώπη. Δεύτερον, δεν έχει μέσο δανειστή ε, στο τελευταίας ευκαιρίας ε, και δεν είχε μέχρι τις ε, οριστικές νομισματικές συναλλαγές, outright monetary transactions. Και δεν έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την δυνατότητα να συντονίσει την δημοσιονομική ή φορολογική πολιτική, δημοσιονομική μόνο πολιτική με τα κράτη-μέλη κάθε κεντρική τράπεζα συζητά τη δημοσιονομική πολιτική με την εκάστοτε κυβέρνηση και καθορίζει την νομισματική πολιτική η εκάστοτε κεντρική τράπεζα όχι υποκείμενη ε, στην κυβέρνηση αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές προοπτικές στο χώρο μέσα στον οποίο ασκεί η νομισματική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια έτσι όπως έχει σχεδιαστεί το σύστημα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, όντω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί νομισματική πολιτική για την Ευρωζώνη, αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εθνική ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Δεν υπάρχει ακόμα ενιαία προσέγγιση. Κάτι έγινε ε, αυτή τη χρονιά και δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλα. Οι εθνικές ρυθμιστικές άρχες ε, αντιμετώπισαν κλασικό παράδειγμα ε, της συλλογικής, ε, περιπτώσεων συλλογικής δράσης. Έχουμε διαρροή κεφαλαίων, διαφυγή κεφαλαίων και οι ρυθμιστικές αρχές στις διάφορες χώρες πώς αντέδρασαν. Την αύξησαν αυτή τη φυγή των κεφαλαίων λέγοντας στις εθνικές τράπεζες ότι πρέπει να μειώσουν την έκθεσή τους στα ομόλογα προβληματικών χωρών. Αυτό ήταν λογικό και αναμενόμενο να συμβεί ε, ενώ από τη μία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενδιαφέρονται για την υγεία του δικού τους εθνικού συστήματος. Το έπραξαν για να τηρήσουν ε, τις υποχρεώσεις τους και λογικό, αλλά με αυτή τους την πράξη καταδίκασαν την Ευρωζώνη σε κρίση. Συν της άλλης, όλες αυτές οι δημοσιονομικές ε, πολιτικές στην Ευρωζώνη υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες που γνωρίζετε, το σύμφωνο σταθερότητας, το no bailout κτλ. κτλ. Θα ήθελα να τονίσω το ότι ε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποδείχθηκε αδύνατο να εφαρμοστεί και αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Σίγουρα επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια. Ωστόσο, η απόσταση που μας χωρίζει από την βιώσιμη νομισματική ένωση παραμένει μεγάλη δεν θα επιληθεί η κρίση του ευρώ μέχρι ότου ή μάλλον πριν διορθωθούν τα λάθη αυτά και όλοι συμφωνούν επί της αρχής, αλλά στη συνέχεια ο καθένας δρά, λες και μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να αναβάλουμε επαόριστον αυτές τις εξελίξεις. Χρειαζόμαστε τραπεζική ένωση, σε κάποιο βαθμό δημοσιονομική ένωση και σε μεγαλύτερο βαθμό πολιτική ένωση. Τραπεζική ένωση τι σημαίνει. Μία εποπτική αρχή, κοινή αρχή για την ε, για το resolution και ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων καταθέσεων. Αυτά, αυτές οι τρεις συνιστώσεις είναι απαραίτητο συστατικό για οποιοδήποτε είδους τραπεζική ένωση έχει υπάρξει ή πρόκειται να υπάρξει ποτέ στην οικονομική ιστορία του κόσμου μας ενιαία εποπτική αρχή, το έχουμε συμφωνήσει. Η διαδικασία όμως για να φτάσουμε μέχρι εκεί είναι τόσο δίσκαμπτη που πραγματικά εξαντλούμε την, ηρεμία, την ε, υπομονή των αγορών. Οι κυβερνήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο ε, ε, ελιγμών. Τα θέματα των stress test, της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών είναι πολύ επικίνδυνα με το κοινό fiscal backstop. Η Common Resolution Authority είναι στο εμβρυϊκό της στάδιο θα έλεγα. Είναι θέμα που είναι υποσυζήτηση και θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία που για μένα έχουν σημασία. Πρώτον, θα εφαρμοστεί ενιαία και με τον ίδιο τρόπο αυτό το οποίο ονομάζουμε η ιεραρχία του ραμφίσματος ως προς τις απώλειες, in order of losses ε, οι απώλειες θα τις επομιστούν ε, ιεραρχικά πρώτον οι πιστωτές, μετά ε, και στο τέλος οι καταθέτες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υποτίθεται ότι έτσι θα ήταν τα πράγματα στην Κύπρο, αλλά τελικά είπαμε και υποτίθεται ότι η Κύπρος θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση που δεν θα ξανασυνέβαινε, αλλά τελικά έχει υποθεί ότι τέτοιου είδους πράγμα μπορεί και να ξανασυμβεί και πώς θα εφαρμόσουν όλους αυτούς τους κανόνες εάν επέλθει κρίση στον τραπεζικό τομέα σε μια συγκεκριμένη χώρα, σε μια οποιαδήποτε χώρα. Από εκεί και πέρα ε, υπάρχει η τάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η Γενική Διεύθυνση της για τον ανταγωνισμό να δρά τρόπον την να, ως η αρχή που θα αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της συγκεκριμένης τράπεζας στην Ευρωζώνη. Καμία τράπεζα στον κόσμο, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει δεχθεί ε, τον ρόλο της ανακεφαλαιοποίησης ε, και του χωρισμού της τράπεζας σε καλή ή κακή ή σε οτιδήποτε άλλο να ανατεθεί ο ρόλος αυτός σε μια γενική διεύθυνση ανταγωνισμού. Ποτέ δεν έχει αποφασιστεί. Είναι πρωτοτυπία παγκόσμια της ε, Ευρωζώνης τον ρόλο αυτό να το αναλάβει μια διεύθυνση ανταγωνισμού. Καμία χώρα ποτέ δεν το έχει διανοηθεί τις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών να τις επιβλέψει και να τις διαχειριστεί μια οποιαδήποτε υπηρεσία ανταγωνισμού της χώρας αυτής. Και βεβαίως λείπει το Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων. Να σας πω τα εξής. Υπάρχουν κάποιες καλές ισπανικές τράπεζες, αν όχι και πολλές. Στο βαθμό που η κατάθεση έστω και ενός ευρώ σε μια καλή ισπανική ε, τράπεζα θεωρείται χειρότερη ποιοτικά σαν στοιχείο ενεργητικού από την κατάθεση του ιδίου ευρώ σε μια κακή γερμανική τράπεζα, όσο αυτή η κατάσταση παραμένει, η, κρίση η ευρωζώνη θα έχει πρόβλημα. Θα έλεγα ότι είναι φυσικό το κίνητρο να φεύγουν τα χρήματα από καλές τράπεζες της περιφέρειας, διότι θεωρούνται τα στοιχεία ενεργητικού εκεί ως ευρισκόμενα εν κινδύνο και θα πηγαίνουν πάντοτε σε τράπεζες του κέντρου της Ευρώπης που θα θεωρούνται πιο ασφαλές. Πάντοτε θα ενισχύεται αυτό το κίνητρο γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο και γιατί είναι και φτηνό. Και όσο ε, παραμένει αυτό, ε, δεν θα αξιολογούνται οι τράπεζες με βάση τα πραγματικά τους βιβλία, αλλά με βάση το fiscal backstop. Και αυτό είναι δυστυχές. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και να, πραγματικά να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινό ταμείο εγγύησης καταθέσεων να ε, μιλήσω λίγο για την Ισπανία στο τέλος της παρέμβασής μου. Ναι, ε, κάναμε πολλά πράγματα εμείς στην Ισπανία που ήταν λάθος. Το ίδιο όμως έκαναν και οι πιστωτές μας. Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα μεταξύ οφηλετών και πιστωτών είναι διμερές το πρόβλημα. Έχουμε αρνητικά επιτόκια πάνω από πέντε χρόνια στην Ισπανία οποιοδήποτε ορθολογικά σκεπτόμενος αναλυτής θα ε, μιλήσει για χρέος που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν είναι βιώσιμο. Το σύστημα που θέσπισε η ΟΝΕ είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζει την μη ορθολογική λήψη αποφάσεων. Εάν δεν εντάξουμε το οικονομικό σκέλος στην νομισματική ένωση, την πραγματική οικονομική ένωση, τότε σίγουρα θα διαλυθεί κάποια στιγμή η Ευρωζώνη και αυτό είναι βέβαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Λάγκε έχει ήδη πάρει το λόγο. Έχουμε τον κύριο Κούλμαν, την κυρία Κλέμπερν, Έμπι, Σάντσεθ Πεσέδο, Λέους, κύριος Χατζηγεωργίου και κυρία Παπαδοπούλου. Μετά από τον κύριο... Α, συγγνώμη, δεν σας είδαμε. Ήμουν πριν από τον κύριο Λάγκερ. Ωραία. Είστε κι εσείς στον κατάλογο. Ο χρόνος ε, μας πιέζει πάρα πολύ. Ακολουθούν δύο πάνελς. Πραγματικά θα το εκτιμούσα αν δεν μιλούσατε για περισσότερο από δύο λεπτά. Ο κύριος Μπούλβαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ο καθηγητής ε, Ζωριών έχει αναλύσει τις ε, δυνάμεις που κινούν το χρήμα μες στην Ευρωζώνη, ενώ ο κύριος Φερνάντες αντιμετώπισε το θέμα της ε, ενδεχόμενης κατάρρευσης της Ευρωζώνης. Θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της Ευρωζώνης έχουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την κρίση. Η μία διάσκεψη κορυφής ακολουθεί την άλλη μετά από το φθινόπωρο του 2009, αλλά δεν έχουμε βγει ακόμα από το τούνελ. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αυτή η αλληλουχία των διασκέψεων κορυφής. Γυρίστε πίσω αν θέλετε στο φθινόπωρο του 2009 και πέστε μας. Πώς κρίνετε τις πολιτικές αντιδράσεις των κρατών μελών. Έδρασαν εγκαίρως, έδρασαν προς τη σωστή κατεύθυνση ή θεωρείτε όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήταν πολύ καθυστερημένη η θεωρειται οπως το ευρωπαικο κοινοβουλιο οτι ηταν πολυ καθυστερημενη η αντιδραση τους και κατόπιν εορτής. Και αν δεν το έκαναν αυτό το 2009, το 2010 παραγωγός στην περίπτωση της Ελλάδος η κρίση είχε κλιμακωθεί στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια το τελευταίο σημείο η λεγόμενη Τρόικα με το απρόσωπο αυτό πρόσωπο που έχει, που έχει λάβει αποφάσεις στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι καθόλου υπόλογη σε κανένα. Ήταν το κατάλληλο εργαλείο για να αντιμετωπιστεί η κρίση της Ευρωσόνης. Ή θα χρειαζόταν περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος, περισσότερη υποστήριξη και δημοκρατική νομιμοποίηση που συμπεριλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης. Ευχαριστώ κύριε Βούλμαν. Ο κύριο Λάγκερ νομίζω ότι θέλει να προσθέσει κάτι σε ό,τι αφορά το δεύτερο μιλητή. Θα ήθελα να ε, εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για αυτά που είπε ο δεύτερος ομιλητής. Υπάρχει το πολιτικό εγχείρημα του ευρώ, το οποίο θα οδηγούσε σε πιο στενή ε, σε πιο στενό συνονισμό και καλύτερη λειτουργία των δημοσιονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είχα ποτέ αμφιβολία ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει γίνει ήδη. Αλλά είπε ο καθηγητής ε, Φερνάντες ότι δεν λειτουργήσε η... το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κάτι μέλη το υπέγραψαν, μετά όμως το έγραψαν, δεν έκαναν τίποτα για να το εφαρμόσουμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή την κατάσταση, την προβληματική που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά μέχρι να ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν είναι αποτέλεσμα εσωτερικών σφαλμάτων, ήταν αποτέλεσμα των, ε, της χρηματοπιστωτικής κρίσης όταν έφτασαν τα παράγωγα να είναι όχι μόνο τρεις φορές η παγκόσμια οικονομία, αλλά 12 φορές η παγκόσμια οικονομία το 2007. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να υπάρχει στάθμιση μηδενική σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο των κρατικών χρεών. Επομένως υπήρξαν πολλά εσωγενή σφάλματα στο σύστημα αυτό. Ναι, έγιναν σφάλματα, όλοι έχουμε κάνει σφάλματα, αλλά τα πράγματα δεν θα ήταν διαφορετικά αν υπήρχε ο δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ θα πρέπει να διαφωνήσω με τον κύριο Μπούλμαν. Είναι θέμα των κρατών μελών να εξασφαλίσουν το δικό του καθήκον και το ερώτημα μου για αυτό του δύο καθηγητέ είναι τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχαν κάνει οι χώρες του Νότου της Ευρώπης για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Ο κύριος Λάμπερς για δύο λεπτά. Αργότερα. Α. Λέβα. Ευχαριστώ, za Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Θα πρέπει να μιλήσουμε σήμερα για συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν το τι ακριβώς έκανε η, η Τρόικα και ποια είναι τα προγραμματά της. Η Τρόικα δεν έχει πάει στη Σλοβενία. Η Τρόικα δεν έχει πάει ακόμα στη Σλοβενία και δεν έχουμε ζητήσει την αρρωγή της. Αλλά είδαμε να γίνονται διάφορες ενέργειες στη Σλοβενία τις προηγούμενες εβδομάδες και κυρίως μέσα στα πλαίσια των δοκιμασιών αντοχής των stress test του τραπεζικού συστήματος Γίνονται αυτές οι δοκιμασίες τώρα σε οκτώ τράπεζες και παραμένουν πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη μεθοδολογία που έχει ακολουθήσει η Κομισιόν και θα πρέπει να εφαρμόσει σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση και τις δοκιμασίες αντοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν έχετε κάποια άποψη σχετικά με τα stress test αυτά καθώς και τη μεθοδολογία που είναι θέμα προσυζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, τι είδου ε, μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί για να έχουν ένα θεμητό, ένα νόμιμο αποτέλεσμα αυτά τα stress test. Η Σλοβενία πολύ φοβάται ότι θα γίνει το πειραματόζωο αυτών των διαδικασιών. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν το Δεκέμβριο και θα ήμασταν πραγματικά ευγνώμονε αν είχαμε κάποιο σχολιασμό από μέρου σα. Ευχαριστώ. Κύριο Σέμπιν. Oh, he disappeared. Sorry. Α, εξαφανίστηκε. Ο, ο κύριος Σάντσεπ Σέντο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ, παρόλο που κάθε κρίση είναι διαφορετική, γιατί δεν είναι το ίδιο αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με αυτό που συνέβη στην Πορτογαλία και με αυτό που συνέβη στην Ιρλανδία και με αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία και στην Ισπανία. Ωστόσο υπάρχει κάτι που αγγίζει όλες τις κρίσεις και το οποίο είναι ότι η νομισματική ε, πολιτική ε, ενδεχομένως ε, ε, βοηθά περισσότερο τις χώρες του κέντρου παρά τις περιφέρειες, λόγω των ανισορροπιών στο σύστημα και λόγω του ότι βεβαίως υπάρχει και έλλειμμα διακυβέρνησης. Εμείς ανέκαθεν ζητούσαμε πολιτική δημοσιονομικής ενοποίησης, όχι τόσο στο άμεσο μέλλον, αλλά με σκοπό να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και να έχουμε συνολικό χρέος μικρότερο σε επίπεδο Ευρώπης. Ναι, αυξήθηκε το κρατικό χρέος και μειώνεται το ιδιωτικό. Όμως στην περίπτωσή μας ήταν το αντίθετο. Στην περίπτωση της Ισπανίας το ιδιωτικό χρέος ήταν τεράστιο και αυτό ε, οδήγησε στην αύξηση του δημοσίου χρέους. Είχαμε βραχυπρόθεσμα δάνεια που συνήφθησαν για ε, το στεγαστικό κλάδο. Δεν είχε υψηλό χρέος η χώρα μας. Το ιδιωτικό χρέος ήταν μεγάλο και τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αναλαμβάνει τους κινδύνους είναι αυτή που ε, μετακυλεί το λογαριασμό στον Ισπανό φορολογούμενο. Και έτσι το εσωτερικό ιδιωτικό χρέος μετατράπηκε το εξωτερικό μάλλον ιδιωτικό χρέος μετατράπηκε σε εσωτερικό εθνικό κρατικό χρέος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κοινή ερμηνεία της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται να την πληρώνουν πάντοτε οι αθώοι. Θα πρέπει και αυτοί που δεν μερίμνησαν και δεν προφυλάχθηκαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς είμαστε υπέρ της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης. Δεν συνέβη αυτό στην Ισπανία. Αν αναλύσει κανείς τη διαχείριση της ε, ε, κρίσης, σίγουρα πιστεύει ότι το να μην επιμένει κανείς στην άμεση ανακεφαλαιοποίηση είναι λάθος. Ευχαριστώ, Αντώνη, λέει ο Πρόεδρο. Για δύο λεπτά ο κύριο Σοφοκλέους, παρακαλώ. Καταρχά Καταρχάς, πλέον προσφέρουμε καλή υπηρεσία εάν παραδεχτούμε ότι η πολιτική και οι αποφάσεις της Τρόικας ήταν και είναι απαράδεκτες, πολιτικά και νομικά ανομιμοποιητές. Δεν υπήρξε πρώτα-πρώτα καμία αλληλεγγύη έβαλε σε περιπέτεια ολόκληρη την Ευρωζώνη. Συμπεριφέρθηκε εκδικητικά στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες και βέβαια συμπεριφέρθηκε ως πειραματόζω όπως εύστοχα έχει λεχθεί σε όλους τους λαούς του Νότου και όχι μόνο. Βήθησε στην ανεργία, τη φτώχεια, την ύφεση, πολλές χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία μιλούν πλέον από μόνα τους. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 33 εκατομμύρια ανέργους. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας στους τέσσερις σήμερα είναι κάτω από τα όρια της στόχης. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή διαπιστώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ξεπέρασε το 1-3. Τι άλλο πρέπει να πει κανείς παρά να παραδεχτεί δημόσια ότι απέτυχε αυτή η πολιτική της λιτότητας. Ίσως πρέπει να ακούσουμε και άλλες φωνές πλέον και νομίζω ότι είναι τεράστια η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην βάλει σε ένα φρένο και να μην συγκρουστεί πολιτικά με αυτή την πολιτική. Ο Κρούκμαν, και κλείνω με αυτό, κορυφαίος οικονομολόγος νομπελίστας σήμερα, στέλνει ένα μήνυμα προς όλους και σε εμάς σε αυτή την αίθουσα ότι επιτέλους αυτά που κάνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα από οικονομικής πλευράς ότι πρέπει να περάσουμε πλέον στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη τώρα από τη λιτότητα πρέπει να ξοδεύσουμε χρήματα. μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε επαναλαμβάνω από την ύφεση και να περάσουμε πλέον στην ανάπτυξη. Ας ακούσουμε και μια άλλη οικονομική σχολή που δεν την ακούσαμε για πολλά χρόνια, κυρίως τον τελευταίο καιρό περισσότερο. Thank you very much. Ευχαριστώ, πολύ, κύριε Σοφοκλέους. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. La señora Χάτι Γεωργίου. señora. Ε, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο μέρος με έχει καλύψει ο συνάδελφος αλλά θέλω να προσθέσω αν έχετε καλοσύνη μερικά πράγματα που ασφαλώς πρέπει να αφορούν και τη χώρα από την οποία προέρχομαι που είναι η Κύπρος όπου μία απόφαση καταστροφική για την οικονομία της Κύπρου πάρθηκε από ένα παράνομο όργανο. Το τραγικό όμως στην υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει κανείς να σου απαντήσει. Ούτε σε αυτήν την αίθουσα πιστεύω. Και τώρα θα μου πείτε, «Ε, τα λέω. Δεν υπάρχει κανείς που θα μου απαντήσει. Όταν ρωτήσεις ε, την Κυπριακή κυβέρνηση μα γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση, σου λέει είναι απόφαση της Τρόικας. Αν ρωτήσεις την Τρόικα, σου λέει είναι απόφαση της Κύπρου και της Κυπριακής Κυβέρνησης ε, αυτή η συγκεκριμένη καταστροφική για την οικονομία της Κύπρου, επαναλαμβάνω, απόφαση κουρέματος. Αν ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει είναι αποφάση του διοικητή στην Κύπρο. Και αν ρωτήσει τον διοικητή στην Κύπρο, σου λέει είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας Δεν υπάρχει κανεί να σου πει τίποτα. Και έτσι τα πράγματα είναι τι άλλο από τραγικά. Ένα ερώτημα μόνο. Υπάρχει κανεί επειδή είναι οικονομολόγοι οι άνθρωποι που μίλησαν, με όση γνώση έχουν από την ε, κυπριακή οικονομία μετά το κούρεμα, με δεδομένο ότι δεν μπορεί κανείς να διακινήσει χρήμα, οι τράπεζες ουσιαστικά δεν υπάρχουν, είναι τράπεζες του 1700 κάτι. Ε, όταν χαλάσει η μηχανή του αυτοκινήτου σου, κατεβαίνεις κάτω και με τα πόδια. Αυτό είναι που έχει συμβεί στην κυπριακή οικονομία. Έτρεχε το όχημα με 200 και πάμε με τα πόδια. Υπάρχει κανείς οικονομολόγος που μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτητα, να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας ή κοροϊδευόμαστε όλοι. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Ο κύριος ε, Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Εγώ προέρχομαι μια χώρα εκτός της Ευρωζώνης και μια χαρά τα πάμε και ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να πάρω μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ πάντως θα το κάνω γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το να ξαναγραφτεί η ιστορία και πιστεύω ότι και οι ακαδημικοί θα πρέπει να δώσουν μια εναλλακτική εικόνα. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν ήμασταν στο ευρώ. Προερχόμενος από μια χώρα που το ε, τη δεκαετία του 90 αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα από τα οποία όμως έμαθε. Θα πρέπει να πω ότι με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι θα πρέπει ορισμένες χώρες να φύγουν και αυτό θα τους κάνει για καλό. Πολύ το αμφιβάλλω. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσατε να το σχολιάσετε. Αν θα ήταν καλύτερο να έχουμε περισσότερα παρά λιγότερα νομίσματα στην Ευρώπη. Επίσης ε, θα ήθελα να ζητήσω τη συμβουλή σας. Εγώ σαφώς είμαι υπέρ του να ενταχθεί η Σουηδία στην Ευρωζώνη. Νιώθω μία μικρή μοναξιά θα έλεγα. Μήπως θα μπορούσατε να με συμβουλεύσατε τι θα μπορούσα να πω στους συμπολίτε μου. Για ποιο λόγο κάνει καλό το ευρώ στην Ευρώπη και πραγματικά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο σε μερικού μήνε θα ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ η Λετωνία. Ευχαριστώ. Τέλος θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λίαμ Όνιοκ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πολ Ζωριών για την ποιότητα της παρουσίασής του, αλλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Αν δούμε τα στοιχεία, <clears throat> τα αριθμητικά, βλέπουμε στις χώρες που είναι υπό πρόγραμμα διάσωσης, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν οδήγησαν σε μια μείωση των ελλημάτων, μεν, αλλά παράλληλα υπήρξε αύξηση της, ε, του ποσοστού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Επομένως, με παράδοξο τρόπο, η προσπάθεια περιστολής του χρέους οδηγεί σε μεγαλύτερη υπερχρέωση. Μία από τις λύσεις που προτείνει λοιπόν ο κατηγητής Ζωριών σημαίνει ουσιαστικά αναδιάρθρωση του χρέους. Το ερώτημα μου το εξή. Για τις χώρες αυτές που βρίσκονται σε μνημόνιο, σε βοήθεια, τι ύψος αναδιάρθρωσης του χρέους κατά την εκτίμησή του είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Excuse me, I made a mistake. Uh, uh, thank you. Συγγνώμη, έκανα ένα λάθος. Ευχαριστώ, κύριε ε, Λία Μιόγκ. Θα ήθελα να πάω εδώ στο λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου, πριν από εσάς. Okay. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα προσεκτικά τι έχει πει ο δεύτερος ομιλητής και θα συμφωνήσω απόλυτα. Λάθος ο σχεδιασμός της ΟΝΕ, απροετοίμαστη η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει κρίσεις, πραγματικά ελλειπής η νομισματική πολιτική δεν ήταν ενιαία και το σύμφωνο σταθερότητας δεν λειτουργήσε το αποτέλεσμα είναι μια πρωτότυπη άδικη λύση από το eurogroup στη δική μου χώρα την κύπρο. δεν μπορεί άγρια ξημερώματα να αποφασίζει το eurogroup και ο κύριος ντάουζεμπλουμ ενώ ο κύριος γιούγκερ είπε όταν ήταν ο ίδιος πρόεδρος του eurogroup δεν θα χρησιμοποιούσε τους κύπριους ως γκάγκστερς. δυστυχώς το eurogroup χρησιμοποίησε την κύπρο και το λαό της ως πειραματόζωα και αυτό το στυλιτεύουμε γιατί σήμερα υπάρχει ανεργία υπάρχει κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι πολιτικέ λιτότητα στην κύπρο απέτυχαν παταγωδώς και θα πω ότι ναι η τρόικα δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση υπάρχει έλλειψη διαφάνεια, δεν υπάρχει αρχή τη λογοδοσία και δεν υπάρχει έλεγχο. ούτε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ούτε από εθνικά κοινοβούλια. και η ερώτηση μου είναι ξεκάθαρη γιατί στην περίπτωση τη κύπρου δεν έγινε κούρεμα χρέου και έγινε κούρεμα κατά τι μπορεί να γίνει τώρα. Εγώ ζητώ και για τη χώρα μου κούρεμα χρέου. όπως έγινε στην Ελλάδα, όπως έγινε και σε άλλες χώρες. Και η ερώτηση μου είναι η εξή: Όταν συζητούμε εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο παραδέχτηκε λάθη. Το λάθος στον πολλαπλασιαστή που έγινε στην Ελλάδα το λάθο για τι άδικε αποφάσει του Eurogroup. Εγώ θα πω στου Γερμανού συναδέρφους ότι κάναμε και εμεί τα δικά μα λάθη. Ε, Μπορούσε η Κύπρος πολλέ μεταρρυθμίσεις να τι είχαμε κάνει από μόνοι μας. Αλλά ο τρόπο που μα συμπεριφέρθηκαν ω Ευρωπαίου πολίτε, θεωρώ ότι ήταν άδικος και δεν έδειξαν κοινοτική αλληλεγγύη. Τι ιδέων γενέστε σήμερα Παίρνω το λόγο για ένα θέμα διαδικαστικό. Έχουμε καλέσει αξιόλογους ε, επιστήμονες εδώ εδώ γίνεται μία συζήτηση μεταξύ βουλευτών που μιλάνε για το πρόβλημα της Ελλάδας, Κίνου κτλ. Τι λόγο είχαμε να καλέσουμε όλους αυτούς, όλες αυτές τις προσωπικότητες. Ξέρετε την άποψή μου για την ακρόαση. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε λόγο στους ειδικού να μιλήσουν. Μίλησαν και μετά παίρνουν το λόγο οι βουλευτές. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μια τάξη εδώ. Είπαμε ότι καλέσαμε προσωπικότητες, θα πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ας τους αφήσουμε το χρόνο να απαντήσουν όπως πρέπει. I think point was... Νομίζω ότι έχει δίκιο. Θα επανέλθουμε τώρα στους ειδικού για να δώσουν τις απαντήσεις τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν αυτό που θέλετε να πείτε το, το έχει ήδη πει κάποιο άλλο, δεν χρειάζεται να πάρετε το λόγο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στο καθηγητή Ζώριον. Επιλέξτε ποιος θα πάρει πρώτος το λόγο. Ναι, θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Γκοζές μας θέτετε ερωτήματα, μπορούμε να απαντήσουμε τουλάχιστον μέρη, αλλά δεν θα έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να υπογραμμίσω και το εξή. Πριν από τρία χρόνια είχα ξαναέρθει σε αυτήν εδώ την αίθουσα και σας απίφθηνα το λόγο ε, στην αρχή της κρίσης που άρχισε τότε να πλήττει την Ελλάδα προτάθηκαν λύσεις σε αυτήν εδώ την αίθουσα για το τι θα έπρεπε να γίνει. Σήμερα ε, βλέπουμε ότι όντως έπρεπε να είχαν γίνει αυτά τα πράγματα και δεν έγιναν. Άρα τίθεται το ερώτημα της εξουσίας που έχει ε, αυτό το όργανο, το, αυτό το θεσμικό όργανο. Η λιτότητα ήταν η χειρότερη λύση και αυτή η λύση είναι που πράγματι υιοθετήθηκε από την Τρόικα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι ε, ε, τα τρία μέρη της Τρόικα κινητοποιούνται με βάση την ίδια ιδεολογία, την συμμερίζονται όλη αυτή την οδολογία, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα στοιχεία, τα αντικειμενικά στοιχεία. Βασίζουν τις αποφάσεις τους σε μια οικονομική θεωρία η οποία διατυπώθηκε για ιδεολογικούς ε, λόγους και η οποία δεν έχει σχέση με την επιστημονική μεθοδολογία. Στρέφουμε τώρα στον κύριο Λάγκε και λέω το εξής. Το ερώτημα επιλύεται με βάση τους όρους που έχουν υπάρξει στη διατύπωση του ερωτήματος. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Η λύση δεν θα δοθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο, γιατί το πλαίσιο ε, είναι κατά τη γνώμη μου το προβληματικό και το είπε και ο κύριος Φερνάντες και το έδειξα. Ίσως μίλησα πολύ γρήγορα. Ε, μίλησα για τα επιτόκια και το έδειξα, αυτό το απέδειξα ότι το σύστημα είναι προβληματικό. Και ο, ο καθηγητής Hans Werner Zinn αλλά και ο κύριος Τίμορ Βολοχόιζερ ε, το έχουν αποδείξει αυτό, έχουν προσεγγίσει αυτό το ερώτημα με διαφορετικούς όρους και χρησιμοποιούν τα στοιχεία στόχου 2, target 2, και έχουν καταλήξει στο ίδιο επιστημονικό συμπέρασμα το οποίο θα συνοψίσω σε μία πρόταση ως εξής. Είναι φερέγγια η Ευρωζώνη και παραμένει φερέγγια, άρα η κατάσταση παραμένει ασταθής και ευπαθής ή θα μειώσουμε το μέγεθος της Ευρωζώνης για να περιλάβει μόνο τις φερέγγιες χώρες ή θα παραμείνουμε ε, ε έχουμε από πλευράς αριθμού μελών Ευρωζώνης και θα υπάρξει ε, ε, συνολική στάση πληρωμών για καθάριση και εξυγίαση της Ευρωζώνης ώστε να καταστεί φερέγγια στη συνέχεια. Και ο κύριος Βούλβες Χόιζερ και ο κύριος Ζιν το έχουν μελετήσει το θέμα. Από τις 17 χώρες ε, της Ευρωζώνης μόνο τέσσερις δεν βιώνουν κρίση. Φιλανδία, κατά χώρες, Λουξεμβούργο και Γερμανία. Όλες οι άλλες χώρες βιώνουν κρίση. 13 από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης. Ξέρω ότι έχετε άλλα στοιχεία εσείς και διαφορετικά, εκτός μικροφώνου ο κύριος Λάγκη. Α, ναι, και η Αυστρία, συγγνώμη. Και το Βέλγιο βιώνει κρίση και η Αυστρία δεν είναι ότι δεν βιώνει κρίση, σε οριακό επίπεδο βρίσκεται και η Γαλλία είναι κάπως στο κόκκινο. Κοιτάξτε, παρακαλώ να εξετάσετε τα αριθμητικά στοιχεία από το στόχο 2. Μόνο 4 χώρες ε, ε, είναι στο πράσινο και 13 χώρες είναι πραγματικά στο κόκκινο οι δείκτες τους. Η Πρόεδρος, δεν χρειαζόμαστε βουλευτές για να κάνουν τη συζήτηση πιο ε, ενδιαφέρουσα. Να δώσω το λόγο στον Φερνάντο. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θα είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μου έχετε θέσει, ε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Να υπογραμμίσω τα πιο σημαντικά σχόλια κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, να μην συγχαίουμε τις χώρες που έχουν ε, έλλειμμα πληρωμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα βιώνουν κρίση το target του, ε, ε, ο στόχος 2 αντικατοπτρίζει τη θέση του ισοσυγείου πληρωμών και του ελλείμματος. Ναι, βεβαίω υπάρχει παρατεταμένο έλλειμμα και οι χώρε αυτέ θα πάνε καλά και από πλευρά οικονομική ανάπτυξη και από πλευρά δημιουργία θέσεων απασχόληση και ικανότητα εξυπηρέτηση του χρέου. Δεν είναι το ίδιο αυτά τα δύο. Από εκεί και πέρα. Το θέμα τη αλληλεγγύη είναι σημαντικό. Βασική μου παρατήρηση είναι η εξή. Δεν είναι κρίση λόγω αλληλεγγύη, είναι κρίση γιατί δεν έχουμε μια λειτουργική οικονομική και νομισματική ε, ένωση. Η αλληλεγγύη είναι ε, μία αγαπημένη λέξη για πολλούς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει οι ΟΝΕ να είναι μια νομισματική ζώνη η οποία να είναι βιώσιμη. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμη γιατί δεν έχει τα βασικά συστατικά που έχει οποιαδήποτε νομισματική ένωση στον κόσμο. Μια κεντρική τράπεζα που να μπορεί να κάνει νομισματική πολιτική για το σύνολο της ζώνης, μια τραπεζική ένωση, που ένα τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί ως ένα και όχι κατακαιρματισμένο, να τη χάνουν ίσης αντιμετώπισης όλες οι τράπεζες στην Ένωση από την ίδια ρυθμιστική αρχή, από τον ίδιο επόπτη και από την ίδια αρχή για τη διάλυση ή ρευστοποίηση ή εξυγίανσή τους και θα μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια πραγματικά βιώσιμη τραπεζική ένωση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγγιήσεις Καταθέσεων δεν είναι για λόγους αλληλεγγύης που θα γίνει. Είναι γιατί είναι βασική προϋπόθεση για να υπάρχει ένα νόμισμα σε μια ζώνη και αυτό έχει φανεί στην παγκόσμια οικονομική ιστορία από την αρχή της μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα. Δεν έχω δει κρίση υπερβολικού χρέους που να μην έχει ε, επιληθεί μέσω της λιτότητας. Όντως χρειάζεται εξυγίανση δημοσιονομική για να μπορεί κανείς να ανασυγκροτηθεί ως χώρα, ως οτιδήποτε για να αποπληρώσει τους ε, ε, πιστωτές του. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την λιτότητα σε κάποιο βαθμό. Τα επίπεδα του χρέους, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, δεν θα είναι βιώσιμα. Έχουμε το εξαιρετικό προνόμιο το εξή. Τα περισσότερα αναδυόμενα κράτη του κόσμου συνεχίζουν να πιστεύουν πιστεύουν ότι το καλύτερο ε, ε, που μπορούν να κάνουν με τα χρήματά τους είναι να τα δώσουν σε εμά για να συνεχίσουμε να συντηρούμε το κράτος πρόνοιας που έχουμε. Αυτό δεν θα το πιστεύουν για πολύ. Κάποια στιγμή θα τελειώσει ε, το χρέος, των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά υψηλό. Μόνο θα μειωθεί από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Ε, η κρίση περιπλέκει όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι όμως αυτά στη ρίζα. Ε, ε, δεν είναι όμως όλα αυτά τα σχόλια που βρίσκονται στη ρίζα του προβλήματος. Και απευθύνομαι τώρα στον Ισπανό βουλευτή και θα ήθελα να μιλήσω λίγο ισπανικά γιατί όντως πολλά έχουν υποθεί για το, για το ισπανικό ζήτημα. Επιμένω, στην Ισπανία κάναμε κάποια πράγματα αρκετά αν θέλετε που είναι λάθος. Η κρίση όμως είναι αποτέλεσμα μιας ατελούς ονέ. Η Ισπανία διατήρησε δημοσιονομική η πολιτική εξαιρετικά επεκτατική και για πάρα πολλά χρόνια δεν είναι μόνο αληθές ότι το δημόσιο χρέος ήταν στα 100% του ΑΕΠ γιατί μετατράπει σε δημόσιο χρέος το ιδιωτικό χρέος. Το κόστος της ανακεφαλοποίησης ε, των τραπεζών είτε έχουμε στοιχεία από το ΔΝΤ του είτε από την ΕΚΤ ε, ε, ήταν μόνο στο 6,7% ως ποσοστό του συνολικού χρέους. Έχουμε έκτακτα δημοσιονομικά έσοδα λόγω της φούσκας στον ε, κτηματομεσητικό τομέα και τελικά ε, δημιουργήσαμε ένα κράτος πρόνοιας πάρα πολύ γενναιόδωρο, πολύ πιο γενναιόδωρο από ό,τι θα μπορούσε να στηρίξει η Ισπανική οικονομία. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό με την Νομισματική Ένωση. Τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε υιοθετήσει το ευρώ. Δεν θα είχαμε ρυθμό ανάπτυξης 4% για τόσα πολλά χρόνια. Θα είχαμε πολύ λιγότερο ενδεχομένω. Σίγουρα είναι θετικό το εισηγείο της προσχώρησης της Ισπανίας στο ευρώ. Καλώς κάναμε και μπήκαμε στο ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνέβησαν διαδικαστικά λάθη. Και βέβαια συνέβησαν, δεν έγινε σωστή διαχείριση της δημοσιονομικής, οικονομικής πολιτικής στην Ισπανία και έγιναν και λάθη στη διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήθελα να ε, πω κάτι που είχε πει ο Ρωμάνο Πρόντι το 2001 όταν πήρε το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε τα εξή και παραθέτω τα λόγια του. Είμαι πεπισμένο ότι το ευρώ θα μα αναγκάσει να θεσπίσουμε μια νέα σειρά μέσων για την ε, νομισματική πολιτική. Είναι πολιτικώ αδύνατο να τα προτείνουμε σήμερα, εν έτη 2001. Κάποια στιγμή όμω θα προκύψει κρίση και τότε θα υιοτηθούν νέα εργαλεία πολιτική. Έχει έρθει, τέλο τη παράθεση. Έχει έρθει λοιπόν η κρίση και τα εργαλεία πολιτικής δεν αξιοποιούνται, δεν δημιουργούνται αρκετά γρήγορα σίγουρα και αν δεν δράσουμε κάποιος νέος σπουδαίος πολιτικός άνδρας θα έρθει το 2020 και θα δηλώσει ότι εμείς χάσαμε την ευκαιρία εν έτη 2013 να δώσουμε ένα τέλος στην κρίση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τελειώνει το πρώτο πάνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με διακατέστησαν κατά την απουσία μου. Περνάμε τώρα στην επόμενη συνεδρία που κατάσταση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, αντιμετώπισης κοινωνικής διάστασης. Εδώ έχουμε δύο ομιλητές, τον Διευθυντή του Τμήματος Αναλύσεων και Προβλέψεων του ΟΕΦΣΥΗ, τον κύριο Ξαβιέ Τιμπό και τον καθηγητή Ζιλ Σεμπόλ από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο καταρχάς για 10 λεπτά. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. <laughs> Θέλω να αντιμετωπίσω το θέμα της ανάκτησης ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης αλλά λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την κοινωνική διάσταση, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του πάνελ μας. Θα προσπαθήσω να τα πω απλά. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι μια διαδικασία αποπληθωρισμού των ε, ημερομισθείων και μισθών σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης. Υπογραμμίζω ότι προς το παρόν είναι μείωση των μισθών και όχι γενικός αποπληθωρισμός και υπάρχει φυσικά μια διαφορά μεταξύ του αποπληθωρισμού και της συμπίεσης, της μείωσης των μισθών. Αλλά η μείωση των μισθών είναι κάτι το οποίο θα έχει σημαντικά αποτελέσματα και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο. Εάν δεν το πράξουμε, κινδυνεύουμε να παραμείνουμε μέσα στην κρίση αυτή για πολλά χρόνια. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να σας πω είναι ότι υπήρξε κάποια επιτυχία μετά από την κρίση το να, στο να μειωθούν οι ανισομέρειες στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα μόνο η Γαλλία έχει ένα αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και όλες οι χώρες του Νότου ιδίω έχουν καταφέρει να μειώσουν τα ελλείμματα αυτά τα οποία είχαν πριν από την κρίση. Αυτό είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή επιτυχία για την Ευρωζώνη, αλλά φοβάμαι ότι δεν μπορεί να παραμείνει βιώσιμη και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτή τη φαινομενική επιτυχία για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε καλύτερα μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο ροδόχρωους και δεν θα είναι και στο μέλλον. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό να καταγράψουμε είναι ότι οι χώρες που είχαν πλεονάσματα στο ισοζύγιο αυτό ε, διατήρησαν αυτό το πλεόνασμα. Δεν υπήρξε επανεξισορρόπηση στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Απλώς υπήρξε μία τροποποίηση της κατάστασης της χώρες που είχαν ελλείμματα στο ισοζύγιο των τριωξών πληρωμών τους. Στις χώρες αυτές υπήρξε μείωση της συνολικής ζήτησης μέσω των προγραμμάτων λιτότητος. Πιστεύουν ορισμένοι ότι δεν υπήρξε λιτότητα, δεν υπήρξε μια σειρά, δεν υπήρξε μάλλον άλλη δυνατότητα από τα προγράμματα λιτότητα στην Ευρώπη. Αλλά άμα δείτε τη δημοσιονομική αντιμετώπιση ήταν πραγματικά αρνητική από πολλέ απόψει και οι δημοσιονομικοί πολιοπλασιαστές ήταν υψηλοί. Κάτι το οποίο οδήγησε σε μείωση της ζήτησης και μείωση του ΑΕΠ, αύξηση στην ανεργία κτλ. Αυτό είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουν, γίνει, έχουν μειωθεί τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στις περισσότερες χώρες του Νότου. Κάτι το οποίο τώρα είναι εν είναι η διαδικασία μείωσης των μισθών. Αυτή η διαδικασία μείωσης των μισθών ισχύει κυρίω για τι χώρε του Νότου, σε μικρέ χώρε όπω είναι η Ελλάδα, όπω είναι η Πορτογαλία, ακόμα και η Ιρλανδία που δεν είναι χώρα του Νότου βέβαια, βλέπουμε η συνολική ονομαστική μισθή να είναι σε πορεία μείωση. Αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε αυτέ τι χώρε, Να μειώνονται οι ονομαστικοί μισθοί, όχι μόνο οι πραγματικοί. Σε χώρε όπω η Ισπανία, υπήρξε μια πολύ δυναμική αύξηση των μισθών πριν από την κρίση. Ακόμα και στην Ισπανία έχουν σταθεροποιηθεί και μειώνονται οι ονομαστικοί μισθοί μετά το 2009. Είναι σε πτωτική πορεία. Αν προσπαθήσει τώρα κανείς να βρει ένα αίτιο για όλες αυτές τις εξελίξεις, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υπήρξε η αύξηση της ανεργίας. Ανέρχεται συνέχεια η ανεργία και αυτό συμπιέζει προς τα κάτω τους μισθούς. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ενώ θεωρούσαμε ότι οι τιμές και οι μισθοί είναι σε μεγάλο βαθμό άκαμπτοι και δύσκολο να αλλάξουν, όταν υπάρξει μεγάλη ανεργία και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό υπερκαλύπτεται από την πίεση της ανεργίας και μειώνουν μειώνονται οι μισθοί. Εγώ δεν ακολουθώ αυτά τα οποία λέω στο γραπτό μου έγγραφο, συγγνώμη προ του διερμηνείς, αλλά βλέπετε κάποια γραφήματα που μπορείτε να διαβάσετε στο έγγραφο αυτό και μπορείτε να δείτε το γράφημα 3, όπου έχετε το συσχετισμό μεταξύ ανεργία και μείωση των μισθών στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ζώνης, Ευρωζώνης. Τι θα προκύψει λοιπόν από όλα αυτά. Η μείωση των μισθών είναι κάτι που είναι θετικό ή δεν είναι θετικό για την Ευρωζώνη. Ένα θετικό παράγοντα είναι ότι με τη μείωση των μισθών θα υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα των πραγματικών ισοτιμιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με νομισματικά μέσα γιατί υπάρχει ένα μονάχα νόμισμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν υπάρχει ένα ενιαίο νόμισμα ο μόνος τρόπος να επαναξισορροπηθούν όλα αυτά είναι μέσω των διαφορικών πληθωρισμού ή των μισθολογικών διαφορών και βλέπετε ότι αυτή η διαδικασία προχωρά με θετικό τρόπο. Μπορεί λοιπόν να περιμένει κανείς από τη μείωση των μισθών και κάποιο κέρδος ανταγωνιστικότητος και ακόμα και περαιτέρω ανάπτυξη, η οποία εν καιρό θα μειώσει την ανεργία και θα ξαναφέρει τα πράγματα εκεί που θα έπρεπε να είναι. Αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα στην ιστορία που δείχνουν ότι ένα τέτοιο θετικό σενάριο που βασίζεται στη μείωση των ε, μισθών δεν λειτουργεί. Η Ευρώπη στη δεκαετία του 1930, η Ιαπωνία τα τελευταία 20 χρόνια δεν λειτουργούν. Αυτό δεν λειτουργεί καλά μέσα στην Ευρωζώνη, γιατί όταν μια χώρα παίρνει ανταγωνιστικότητα, τότε οδηγεί σε άλλες χώρες τη μείωση των ε, μισθών. Επομένως μειώνεται το κέρδος ανταγωνιστικότητας που μπορεί να αποκτήσει αυτή η χώρα. Το να διαχέεται με αυτόν τον τρόπο η μείωση των μισθών, αυτό μειώνει την, το κέρδος ανταγωνιστικότητας μέσα στην Ευρωζώνη. Χρειάζονται πραγματικές προσαρμογές εσωτερικής ισοτομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε όλοι θα πρέπει να προσαρμόσουν τις εσωτερικές του ισοτιμίες εναντί της Γερμανίας. Αυτό είναι απαραίτητο και αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτα αλήθεια γιατί ακόμα και στη Γερμανία βλέπει κανείς να υπάρχει μείωση των μισθών. Στο τμήμα τουλάχιστον των χαμηλών αμοιβών, αλλά είναι και εκεί μια διαδικασία μείωση των μισθών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε τι συνέπειε που μπορούν να προκύψουν από μια τέτοια διαδικασία. Το δεύτερο <clears throat> το οποίο μπορεί να αναμένει κανεί από την μείωση των μισθών αυτό είναι λιγότερο σοβαρό από, τον πλήρη αποπληθωρισμό, αλλά σίγουρα η διαδικασία αυτή αυξάνει το βάρος του χρέους για το ιδιωτικό χρέος στις χώρες όπου υπάρχει αυτή η μείωση των μισθών. Το να αυξηθεί λοιπόν το ιδιωτικό χρέος, το βάρο της υπερχρέωσης σε χώρες όπου πρέπει να υπάρξει μια απομόχλευση ε, του ιδιωτικού χρέους και δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, όλα αυτά κάνουν το ιδιωτικό χρέος να είναι ακόμα λιγότερο βιώσιμο. Και ξέρουμε ότι το μη βιώσιμο ιδιωτικό χρέος στο τέλος θα μετατραπεί σε μη βιώσιμο δημόσιο χρέος και το δημόσιο μη βιώσιμο χρέος θα γίνει η αιτία νέων προβλημάτων. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία υπήρξαν στην απαρχή της κρίσης κρατικού χρέους μπορούν να επανέλθουν μέσω της μείωσης των μισθών. Υπάρχει ένα γράφημα το οποίο έχω στο εγγραφό μου, είναι το γράφημα 4, όπου μπορείτε να δείτε τα επισφαλή δάνεια στην Ισπανία και βλέπετε ότι αυξάνονται τα επισφαλή δάνεια ακόμα και μετά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μετά την έκρηξη της κρίσης βλέπετε με αυτόν τον τρόπο ότι η προσαρμογή που γίνεται δεν φέρνει αποτελέσματα. Τρίτον, η συμπίεση των μισθών αυξάνει και την ανισότητα. Στις περισσότερες εργασιακές αγοράς της Ευρώπης υπάρχει μια δυτή αγορά. <clears throat> υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στους χαμηλούς μισθούς από τη μείωση των μισθών από ότι στο ψηλό κομμάτι των μισθών. Περισσότερη πίεση στους μισθούς φυσικά γίνεται από ότι στο εισόδημα από κέρδη κεφαλαίου και άλλες μορφές ε, ε, εισοδημάτων. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αυξάνεται η ανισότητα. Έχουμε ένα παράδειγμα τύπου Στίγλιτς. Ο Στίγλιτς έλεγε ότι η ανισότητα είναι ένα από τα αίτια της κρίσης. Το παραδόξο είναι ότι η κρίση ουσιαστικά αυξάνει από μόνη της την ανισότητα αυτή. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για όλα αυτά. Τι εναλλακτική λύση έχουμε από τις συμπίεση των μισθών και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Σε 20 δευτερόλεπτα λοιπόν θα το πω αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αναχαιριστεί η μείωση της συνελικής ε, ζήτησης. Αν ε, παρατείνουμε στο χρόνο και μειώσουμε τη λιτότητα, γίνεται η ίδια προσαρμογή, αλλά γίνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όχι βραχυπρόθεσμα. Και με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να έχει χαμηλότερους πολλαπλασιαστές. Με χαμηλότερους πολλαπλασιαστές έχει κανείς περισσότερα θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του χρέους και λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στην ανεργία. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν στοιχείο. Επίσης είναι σημαντικό να κοιτάξουμε το μακροπρόθεσμο επίπεδο όταν μιλάμε για την βιωσιμότητα του χρέους. Όταν θέλουμε τη βιωσιμότητα σε σύντομο μονάχα διάστημα καταλήγουμε σε μη βιώσιμο χρέος και έχουμε κάποιες ακόμα, έχω εγώ κάποιες ακόμα προτάσεις. Μία πρόταση <clears throat> να εμποδίσουμε την μείωση των ονομαστικών μισθών στην αγορά εργασίας και αυτό μπορεί να γίνει με το να καθορίσουμε ένα επίπεδο χαμηλότερου μισθού αυτό μπορεί να είναι ένα πολύπλοκο σύστημα γιατί θα εφαρμόζεται σε διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα με διάφορα, διαφορετικά επίπεδα ελάχιστων μισθών, μήνυμου μισθών και να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα για να επιτύχουμε δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε σε κάποιο επίπεδο την μείωση των μισθών. Δεν είναι το, ο πραγματικός φραγμός που θα τα σταματήσει όλα, αλλά μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Και δεύτερον, να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο, ώστε μας σε πρόθεσμα να ξεσορροπήσουμε και πάλι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ώστε οι χώρες που έχουν ε, πλεονάσματα να αυξήσουν περισσότερο το κατώτερο επίπεδο μισθών από ότι η αύξηση της παραγωγικότητάς τους, ενώ οι χώρες που έχουν προβλήματα να έχουν τη δυνατότητα μιας πιο μικρής αύξησης του ελάχιστου μισθού, ενώ ανεβαίνει η παραγωγικότητά τους και έτσι να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ένα τέτοιο εργαλείο λοιπόν μπορεί σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο να αντιμετωπίσει τα θέματα της ανισορροπίας των ε, ισοζυγίων τρέχουσων πληρωμών. Ευχαριστώ. Πολλά ήταν τα 20 δευτερόλεπτά σας. Θα περάσουμε τώρα στο καθηγητή Ζήλ Σεν Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να διαβάσω την εμιλία μου. Οι στόχοι των χωρών που είναι σε φάση προσαρμογής είναι διητοί. Βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να μειώσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης της δημόσιας διοίκησης για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την ε, βιωσιμότητα. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο δυνητικού αποτελέσματος μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η κρίση οδήγησε στην υιοθέτηση μέτρων που προσπαθούν να επιληφθούν και το δύο θεμάτων. Αυτή τη στιγμή αυτέ οι οικονομίε δεν δείχνουν πολλά σημεία βελτίωση. Η ανεργία έφτασε σε ιδιαίτερα κρίσιμα επίπεδα στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η ανάπτυξη παραμένει περιορισμένη και σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά παρόλε τι αργινέ προσπάθειες που έγιναν. Η διαρθρωτική στρατηγική εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο βραχυπρόθεσμα για να, για για αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της προσαρμογής. Η συνολική ζήτηση θα πρέπει να στραφεί προς τις εξαγωγές κάτι που σημαίνει μια υποτίμηση του πραγματικού, των πραγματικών ισοτιμιών. Λόγω του ευρώ αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω μιας υποτίμησης του νομίσματος. Η εναλλακτική λύση είναι μια ελαστικότητα, ε, ελαστικότητα προς τα κάτω των ονομαστικών μισθών, κάτι που σε ορισμένες χώρες, Πορτογαλία για παράδειγμα, δεν φαίνεται να συμβαίνει. Ενώ σε άλλες χώρες είναι μια παρατεταμένη δυσάρεστη διαδικασία η οποία είναι γεμάτη από πολιτικούς κινδύνους. μακροπρόθεσμα για να αυξηθούν τα κίνητρα στην εργασία θα πρέπει κανείς να επανεξετάσει τη γενοδογυρία του κράτους προνοίας. Αυτό όμως αντίκειται στις πολιτικές πλατφόρμες που τα περισσότερα πολιτικά κόμματα πουλούσαν στο εκλογικό σώμα ολόκληρες δεκαετίες. Για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί για την είσοδο στις καλές αγορές. Αυτά τα εμπόδια όμως εξυπηρετούν ορισμένες ομάδες συμφερόντων που είναι κατά της άρσης των περιορισμών. Αυτοί οι περιορισμοί μειώνουν το περιθώριο των ε, αυτών που αποφασίζουν τις πολιτικές και καθιστούν ακόμη πιο σημαντικό την, ε, ε, σημαντική την ανέβρεση ενός διαρθρωτικού πακέτου. Μέχρι στιγμή πιστεύω ότι τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί δεν καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους ιδιαίτερα γιατί η συνοχή μεταξύ των δύο στόχων έχει αγνοηθεί. Έχει αγνοηθεί, όπως είπαμε, αυτή η συνοχή για να μπορούν να επιτύχουν ε, οι διαφορετικέ αυτές προσαρμογές θα πρέπει να αποφύγουμε μέτρα τα οποία ε, εξηγιαίνουν βραχυπρόθεσμα αλλά έχουν αριστικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να αποφύγουμε δεύτερο μεταρρυθμίσεις που οθούν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα μακροπρόθεσμα αλλά έχουν μια άμεση αρνητική επίπτωση οικονομικές δραστηριότητες και στα εισοδήματα από τους φόρους. Η παγίδα του να αγνοούμε αυτές τις προσκλήσεις είναι ότι το πακέτο μεταρρύθμισης θα μπορούσε γενικά να είναι ανεπιτυχές από τη στιγμή που διάφορα σημεία στο όλο πακέτο έχουν αντισταθμιστικές επιπτώσεις και, στη, και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην οικονομία. Επιτρέψτε μου τώρα να αφαιθώ σε ορισμένες πτυχές των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις ε, χώρες που προαναφέραμε υπό το φως αυτό των αρχών. Θα αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα, και το μεταρρύθμιση στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία και θα συζητήσω το βαθμό μέχρι του οποίου υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των επιπτώσεων των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων. Σε ό,τι Μερικέ φορέ ενδεχομένω θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτά και αλλού. Σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική προσαρμογή, τη βράχη πρόθεση θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα μείωση των δαπανών και όχι σε αύξηση του εισοδήματο. Τα τελευταία θα μπορούσαν να συνδυαστούν με μια μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, η οποία έχει αρνητικέ επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει μια γενική συμφωνία σε ό,τι αφορά τα ωφέλη φορολογική συμφωνία πολυμόρφωση, το οποίο αποτελεί μέρο τη μεταρρύθμιση ε, στις, στις παραπάνω χώρε. Πράγματι, καταρχά, μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ίσπραξη φόρων θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα ίσπραξη του ίδιου ποσού με χαμηλότερου φορολογικού συντηρηστέ και με αυτόν τον τρόπο να μειωθούν οι ε, εκτροπέ. ε, αυτό προλύνει το έδαφο για μελλοντικέ αυξήσει από κεροσκοπικέ ε, κυβερνήσει, απλά και μόνο καθιστώντα λιγότερο δαπανηρές αυτέ τι αυξήσει. Στην Πορτογαλία οι αποζημιώσεις καταγγελίας ε, σύμβασης σε εργαζόμενους με μόνιμες συμβάσεις έχουν μειωθεί ε, και με αυτό οδήγησε σε μια ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ η μεταρρύθμιση αυτή ε, θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει και ε, ενώ δίχω άλλο θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα μειώσει την, τη διάρκεια της ανεργία, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναβληθεί. Η άμεση επίπτωση θα είναι να πυροδοτήσει ένα κύμα ε, θέσεων εργασία εν μέσω της ύφεση. Κάτι το οποίο διακυβεύει τους μακροχρόνιους ε, οικονομικούς στόχους μιας χώρας. Κατά τρόπο, η προσπάθεια προσπάθεια να επιβληθούν φόροι στου προσωρινέ συμβάσει στην Ιταλία και στη Γαλλία θα μπορούσε να θεωρηθεί ω ένα χρήσιμο βήμα προ ε, μια, ενοποιημένο, μια ενοποιημένη σύμβαση η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τι ανεπάρκειε του διτού ε, συστήματο. Βράχει πρόθεσμα θα μειώσει τι θέσει εργασία και θα αναβάλει την ε, ανάκαμψη. Από την άλλη πλευρά, η μεταρρύθμιση στον τομέα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Πορτογαλία που μεταξύ των άλλων περιορίζει την αυτόματη η επέκταση των ε, συμφωνιών ε, ως προς έναν ολόκληρο τομέα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτές που συμφωνίες υπογράφονται από συνδικάτα που εκπροσωπούν τη μειοψηφία των εργαζομένων, έχει ωφέλη και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πράγματι, στην Ιταλία έγινε μια παρεμφερής μεταρρύθμιση. Μακροπρόθεσμα θα μειώσει την ισορροπία, ε, το επίπεδο ισορροπίας στην ανεργία ιδιαίτερα από τη στιγμή που ε, ο καταμερισμός εργασίας θα γίνει μέσω των μισθών και όχι μέσω των διαστημάτων ε, του χρόνου ανεργίας. Βραχυπρόθεσμα καθιστά πιο εύκολο να επιτευχθεί το αναγκαίο επίπεδο ρύθμιση των ε, μισθών και να επιστρέψει, επιτρέπει, επιστρέψει σε αποδεκά επίπεδα. Θα, θα, ήθελα να προσθέσω ότι στην περίπτωση της Πορτογαλίας δυστυχώς αυτό θα είναι ανεπαρκές γιατί η απαιτούμενη προσαρμογή στους μισθούς κινείται γύρω στο αφορά μία μείωση κατά 10 ως 20% στις, ε, ονομα, στους μισθούς και αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω μία υποτίμηση η οποία αποκλείεται λόγω του ευρώ. για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι άμεσες επιπτώσεις της κρίσης και ιδιαίτερα το υψηλό ποσοστό ανεργίας, η Ελλάδα επεκτείνει το ε, ε, δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας. Αυτό συμπεριλαμβάνει προσωρινές θέσεις εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση, βασικό εγγυημένο εισόδημα και επέκταση της ε, υγειονομικής περίθαλψης. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά διαθροτικά ταμεία καθώς και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Μολονότι αυτά τα μέσα ε, είναι κατανοητά λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό πλαίσιο δεν είναι συνετά, δεν είναι ορθά. Οι προσωρινές θέσεις εργασίας είναι αποτελεσματικές και προγράμματα όπως το βασικό ελάχιστο μισθό είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταργηθούν και αυξάνουν και θα δημιουργήσουν πραγματικές παδίγες φτώχειας. Η Ελλάδα ενδεχομένω δεν μπορεί να αναχτεί ένα επίπεδο κοινωνικής προστασίας παρεμφερές με αυτό των σκανδιναβικών χωρών. Πιστεύω ότι αυτό μας δείχνει το πώς μια ε, κακή μακρονομική κατάσταση θα μπορούσε να δημιουργήσει δημιουργήσει μια ε, πολιτική, ένα πολιτικό έρισμα για ε, ε, πολιτικές που έχουν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Η άρση των περιορισμών στα προστατευόμενα επαγγέλματα θα πρέπει να έχει θετικέ επιπτώσει και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, ο καταπληκτικό εργασία είναι πιο αποτελεσματικό και το κόστο των υπηρεσιών ε, στου κατανοητέ και στι επιχειρήσει μειώνεται. Βραχυπρόθεσμα, ε, οι άνεργοι θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτά τα επαγγέλματα που ανακουφίζουν το πρόβλημα τη ανεργία. Τελειώνοντα, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου Λόγω της κρίσης οι χώρες εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις που έχουν δύο στόχους. Καταρχάς ε, δημοσιονομική εξυγίαση και μακροπρόθεσμους στόχους προώθηση της ανάπτυξης αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει αφιερωθεί περισσότερη σκέψη για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των μέτρων που ακολουθούνται ε, ε, για να αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα ε, αλλά και τις ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις που υποτίθεται ότι θα είναι αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τον κατάλογο που έχει καταρτήσει η γραμματεία ακολουθώντας τον κανόνα DON'T. Θα σας τους διαβάσω. Αν υπάρχει κάποιος που δεν είναι στον κατάλογο, να μας το πει. Κάποιος άλλος θέλει τον να λάβει το λόγο? Κάποιος άλλος? Βέρνερ Λάγκε. Εντάξει, στο τέλος. Κάποιος άλλος? Κύριος Αλαβράκος. Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω από εδώ. Θα σας περιορίσω σε δύο λεπτά τον καθένα. Παρακαλώ θέστε ερωτήματα και μην κάνετε δηλώσεις. Αλλιώς θα αναγκαστώ να σας διακόψω πρωτού θέσετε το ερώτημα σας. Η Ιβάνα πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίσω το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο σημαντικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κατευθύνει τα κράτη-μέλη και να τα παροτρύνει να κάνουν τις απαραίτητα βήματα για να υπάρχει ανάπτυξη και πλήρης απασχόληση. Αλλά χωρίς να υποσκάψουν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών της. Είναι το ευρωπαϊκό εξάμεινο και η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Συμφωνώ με τους εμπειρογνώμονες ότι είναι σημαντικά τα μέτρα λιτότητος και συμφωνώ μαζί τους ότι πρέπει να έχουν πιο πολύ μεσοπρόθεσμο και όχι βαχυπρόθεσμο χαρακτήρα γιατί οι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα θα πρέπει να βγουν από αυτόν τον φαύλο κύκλο και να ξεκινήσουν την ανάπτυξη και να μειώσουν την ανεργία. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθεί αυτή η κίνηση ώστε να μπορέσουν να βγουν από την κρίση χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα για το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Στο ερώτημα μου λοιπόν προς εμπειρογνώμες είναι πού βρίσκεται η σωστή ισορροπία μεταξύ των μέτρων λιτότητος και της ανάγκης να υπάρξει τόνωση της κατανάλωσης, της ανταγωνιστικότητος και επίσης πώς θα βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και των μέτρων τα οποία δημιουργούν ένα έφορο ε, επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και η εργασιακή δύναμη με πιο εύκαμπτο τρόπο και πώς μπορούν να τροποποιηθούν οι δημοσιονομικές πολιτικές για να μειωθεί η φορολογία στο εισόδημα. Μόνο ένα συνδυασμό αυτών των μέτρων, κατά την άποψή μου, μπορεί να οδηγήσει σε μια αναστροφή των σημερινών τάσεων και να επιλύσει τα προβλήματα, να φέρει ένα πλεόνασμα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά στην πράξη, λοιπόν. Ευχαριστώ. Η Ρώδη Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι σχετική με αυτό που μόλις έκανε συνάδελφος. Ζούμε μόνιμα στην αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ λιτότητας μεταξύ προσαρμογής μέσω λιτότητας και από την άλλη πλευρά την ανάγκη του να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάκαμψης. Θέλω να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες ήδη κατάλαβα ότι υπάρχουν ενστάσεις για το, τα μέσα τους πολλαπλασιαστές που έχουν εφαρμοστεί και για τη διάρκεια της επίτευξης της προσαρμογής της δημοσιονομικής. Θα ήθελα να ρωτήσω, βλέπουν οι ίδιοι και τι θα πρότειναν παράλληλα αν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές έχουν και ένα μακροπρόθεσμο στόχο και μια μακροπρόθεσμη ε, υποδομή για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους οι χώρες μετά το τέλος των προγραμμάτων προσαρμογής ή μετά βρισκόμαστε στο κενό και θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να συζητούμε για το πώς θα επιτευχθεί και η συνοχή και η ισορροπία στην Ευρώπη και η ανάπτυξη αυτών των χωρών. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποδηματά. Το θέμα που συζητάμε σε αυτό το πάνελ είναι αποκαθιστώντας την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, συνυπολογίζοντας τον κοινωνικό παράγοντα, την κοινωνική διάσταση. Στα προγράμματα που εφαρμόζονται εδώ και τρία χρόνια στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα ήταν να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να βαθύνει όμως ταυτοχρόνως σε πολύ μεγάλο βαθμό ύφεση και να αγνοηθεί πλήρως και ο κοινωνικός παράγοντας, η κοινωνική διάσταση, αλλά και ο πολιτικός παράγοντας, ο παράγοντας της πολιτικής σταθερότητας. Και θέλω να ρωτήσω, σας ευχαριστώ και τους δύο καταρχήν για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας. Ο κύριος Τιμπό έκανε δύο παρατηρήσεις που μου φαίνονται ενδιαφέρουσες για την ελληνική περίπτωση. Είπατε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα έπρεπε να είναι τόσο εμπροστοβαρής ή δεν πρέπει να είναι τόσο εμπροστοβαρής αλλά να γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου ώστε και οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές να έχουν μικρότερη επίπτωση στην οικονομία και επίσης ότι το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους θα πρέπει να ε, εξετάζεται πιο μακροπρόθεσμα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή οι παρατηρήσεις σας είναι στον αντίποδα της φιλοσοφίας του ελληνικού προγράμματος, είναι σε λάθος κατεύθυνση το ελληνικό πρόγραμμα, συμμερίζεστε τις εστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα που βελτιώθηκε είναι βιώσιμη αυτή η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με 30% σχεδόν ε, ανεργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κυλακάκης. Κυλακάκης. well, uh, let me, let me, uh, start. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα ερωτήματα και μετά να κάνω την ανάλυση της κατάστασης. Πρώτο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε ε, το ξόδεμα του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Μένουν άνθρωποι άνεργοι 4 και 5 χρόνια. Πόση απασχόληση θα έχουμε μετά από αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Καταστρέφεται ο παραγωγικός ιστός της χώρας για τέσσερα και πέντε χρόνια δεν υπάρχει καμία επένδυση στη χώρα. Γιατί είναι 4 ή 5% η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, της Ελλάδας π.χ. και της Γερμανίας. Έτσι είναι οικονομικός παράλογο να κάνει κανείς οποιαδήποτε επένδυση στην Ελλάδα. Τρίτο ερώτημα. Πώς, ε, ποια είναι η γνώμη σας για την ε, περικοπή των, της πίστοσης σε αυτή την προσπάθεια για να βγούμε από την κρίση. Μπορούμε να έχουμε ανάκαψη της οικονομίας χωρίς πίστοση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μπορεί κανείς να κόψει τα τέσσερα πόδια ενός βατράχου και μετά να απαιτήσει από το βάτραχο να πηδήξει. Δύσκολο κάπως αυτό. Και τέλος, μιλήσατε για τα εισοδήματα. και λέτε ότι αντί να ε, ε, αυξήσουμε την αύξηση των εισοδημάτων, καλύτερα να περικόψουμε τις δαπάνες. Η Τρόικα στη χώρα μας θέλει να αυξηθούν τα έσοδα, το πολιτικό σύστημα το προτιμούσε από τα να μειωθούν οι δαπάνες. Ωστόσο το κράτος ε, δαπανά το 53% του ΑΕΠ ε, ως γενικές κρατικές δαπάνες, περισσότερο και από τη Σουηδία. Το 2012 το κράτος το 50% του ε, ΑΕΠ το δαπανά για γενικές κρατικές δαπάνες. Συνεχίζει δηλαδή. Ποια, πώς ερμηνεύεται αυτή τη διαφορά, να πάμε σε μια προσαρμογή με μικρότερο κράτος ή σε μια προσαρμογή με ε, περισσότερους φόρους. Ευχαριστώ, Φιλίπ Λαμπέρτς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Σαμπόλ. Θα μιλήσω γαλλικά και για να τον ευχαριστήσω και γιατί είναι και πιο εύκολο για μένα. Είστε μηχανικός από ό,τι είδα και στην ε, παρέμβασή σας κάνετε κάποιες δηλώσεις και θα ήθελα ε, να ασχοληθώ με αυτές και να απευθυνθώ κυρίως στην επιστημονική σας πλευρά και όχι τόσο στην τεχνική. Ο συνάδελφος κ. Κυλακάκης μίλησε για το θέμα των εσόδων και των δαπανών είπατε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση των δαπανών, διότι η επιβάρυνση φορολογική ε, ε, διαστρεβλώνει σε βάθος χρόνου την οικονομία και έχει αρνητικό αντίκτυπο. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι σχετικά απλό. Θεωρώ ότι η υπόθεση εργασίας είναι ότι ο κράτος είναι, το κράτος είναι κακός διανεμητής πόρων, ενώ η αγορά είναι καλύτερος. Ποια είναι τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτετε εσείς που στηρίζουν αυτή την τοποθέτηση. Εξ όσων θυμάμαι, η κρίση που γνωρίσαμε το 2008 οφειλόταν κυρίως ε, ε, στην ε, φούσκα ε, των στεγαστικών δανείων στη ΣΥΠΑ, στην Ιρλανδία και αλλού διανέμονται πόροι από τις κυβερνήσεις με αρνητικό, με κακό τρόπο και ο ιδιωτικός τομέας δεν απαλλάσσεται των ευθυνών που έχει και των λαθών που έχει κάνει σε αυτή την κατανομή των πόρων. Ε, επομένως για να είστε τόσο κατηγορηματικό, σίγουρα θα έχετε ε, στέρεα επιστημονική βάση που θα στηρίζει την θέση σας. Ποια είναι αυτή. Δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με την αγορά εργασίας. Είστε μηχανικός και εγώ το ίδιο. Μου αρέσει να παρατείνω τις καμπύλες αν θέλετε. Και αν σας κατάλαβα ε, καλά, κάνουμε μείωση μισθών, όπως την είπε ο κύριος Ταμπό, ε, μειώνουμε τους ονομαστικούς μισθούς ή μειώνουμε την κοινωνική προστασία και έτσι, μειώνοντας όλα αυτά, μειώνουμε και την ανεργία. Έστω, ας πούμε ότι έτσι ισχύει. Εάν σας κατάλαβα καλά, λοιπόν, να συνεχίσουμε με αυτή την άγουσα και σε βάθος χρόνου, σε μια οικονομία όπου το 100% ε, των ανθρώπων θα ήταν δούλοι, τότε θα είχαμε μηδέν ανεργία. Έτσι δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική δήλωση, δικιά μας δουλειά είναι αυτή. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτεται, που επαληθεύουν και επιβεβαιώνουν τις ε, δηλώσεις που μας κάνετε εδώ. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, καλώς, η κυρία Γκόμες τώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον καθηγητή κύριο Σαμπόλ. Ε, και θα ήθελα να μιλήσω για μια έκθεση που δημοσιεύθηκε χθε στην Πορτογαλία και η οποία λέει ότι ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που βασίζεται στην ε, καταβαράθρωση της απασχόλησης και στην ε, εξαφλίωση των μισθών δεν μπορεί να είναι επιτυχημένο. Δεν έχουν τελματώσει, βαλτώσει οι μισθοί στην Πορτογαλία. Καταβαραθρώνονται. Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας μας λέει ότι ο βασικός μισθός είναι 485 ευρώ στην Πορτογαλία και με πραγματικούς όρους μειώθηκε κατά 4,7% κατά μέσο όρο τα τελευταία δύο χρόνια. Συντάξεις ε, της τάξης των 600 ευρώ και πάνω έχουν μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ας πούμε ένα, ένας διπλωμάτης, 40 χρόνια πρέσβης, παίρνει μισθό 3.000 ευρώ το 2011 και σήμερα έχει μισθό 2.500 ε, ευρώ, μια μείωση 20%. Αυτό δεν αυξάνει την παραγωγικότητα, δεν αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, δεν ενισχύει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αυξάνει το κίνδυνο της παιδικής φτώχειας, καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό, την κοινωνική προστασία και ενισχύει την μετανάστευση αφού οι νέοι εγκαταλείπουν την χώρα. Βάσει της έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τα τελευταία χρόνια μία στις 7 θέσεις απασχόληση έχει ε, εξαφανιστεί στην, στην Πορτογαλία. Το 10% έχει εξαφανιστεί από πλευράς θέσεων εργασίας. Οι νέοι, οι πιο προσοντούχοι φεύγουν κάθε μήνα ε, σειραίων στο εξωτερικό, εγκαταλείπουν τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οξύνονται οι ανισότητες, εγκαταλείπουν οι νέοι τη χώρα, έχουμε υψηλή μετανάστευση προς τα έξω, η παρουσία μας στην Ευρώπη πραγματικά υπονομεύεται. Η Πρόεδρος, δεν κατάλαβα ποιο είναι το ερώτημά σας. Συμβάσεις ο κύριος Οάνγκ Γκόγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, ένα ερώτημα για καθένα από τους εμπειρογνώμονες εγώ Είδα πολύ ενδιαφέρον το, αυτό που είπε ο κύριος ε, Τιμπό για τα αρνητικά αποτελέσματα της μείωσης των μισθών. Εμείς στο εκλογικό μας πρόγραμμα θέλαμε να πούμε αυτό το πράγμα, ότι να υπάρχει μία αύξηση των μισθών. Αν μας έλεγαν όμως μετά οι επιχειρήσεις ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε μας. Επειδή βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας το ερώτημα είναι μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια αναθέρμανση των μισθών χωρίς να μειώσουμε το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό στην πραγματικότητα. Στον κύριο Πόλε. μια ακόμα απόχρωση σε αυτά που είπε ο κύριος ε, ε, Λαμπέρ. Πόσο αποτελεσματική είναι η μείωση των δαπανών. Αυτό προϋποθέτει ότι ο πολλαπλασιαστής είναι κοντά στο μηδέν και επίσης ότι ισχύει η ισοδυναμία του Ρικάρντο. Μα μπορώ να σας... Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν να ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά τα δύο, αυτές οι δύο προϋποθέσεις που αναφέρατε. Ο Γιώργιν Κλούτε. Σε ευχαριστώ Σάρον. Πρέπει τα οικονομικά θέματα να μπουν στο προσκήνιο. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω ότι τα μέτρα τα οποία ελήφθηκαν μέχρι τώρα για την ε, αντιμετώπιση της κρίσης είχαν τεράστιες πολιτικές συνέπειες. Υπάρχουν κάποια κόμματα αντιευρωπαϊκά που θέλουν να, διατηρήσουν, να, να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πάρει μεγάλη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να, θέσω ένα ερώτημα τώρα στον κύριο Τιμπό. Μιλάτε για την ανταγωνιστικότητα, αλλά όλα αυτά μου φαίνεται ότι είναι κάπως αφηρημένα. Ήμουνα πρόσφατα στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και είδα κάποια πράγματα τα οποία δεν ταιριάσουν με αυτή την αφηρημένη έννοια της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτές τις χώρες υπάρχει μια σημαντική αποβιομηχανοποίηση. Όταν δεν υπάρχει μια τέτοια βιομηχανία, πώς μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικότητα στην βιομηχανία τους, όταν πρέπει να την ξαναφτιάξουν από την αρχή. Όταν δεν υπάρχει πια παραγωγική βάση, πώς θα μπορέσουν να αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες. Επίσης υπάρχουν πολλές ε, αγροτικές επιχειρήσεις και στις δύο χώρες και στην Κύπρο ισχύει αυτό το πράγμα που δεν έχουν καμία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά γιατί οι μονάδες αυτές παραγωγής είναι πολύ μικρές και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες ε, αγροτοτροφημικές μονάδες. Είναι έτσι ή όχι. Και υπάρχει, υπάρχει και ένας αριθμός χωρών που παράγουν πολύ λίγο για την αγορά τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ε, διαρθρώσεις της παραγωγής ώστε οι χώρες αυτές να έχουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά τους και θα ήθελα να έχω τη δική σας άποψη. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς όλα αυτά τα προβλήματα. Ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά. Ευχαριστώ λέει Σάρον. Ο Νίκ Γκρίφιν. Ευχαριστώ δύο ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε σήμερα το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα ότι η υπενθύμηση που έγινε στο πρώτο πάνελ ότι η κρίση αυτή είναι μια τεχνητή κρίση η οποία έχει δημιουργηθεί από την αρχή σαν πρόσχημα για να υπάρξει μια ε, πολιτική ένωση στην Ευρώπη με την κοινική δήλωση του πρώτη και δεύτερον το θέμα της μείωσης των μισθών στην Νότια Ευρώπη. Ακούγοντας αυτά που είπαν, βλέπω το ίδιο πράγμα να γίνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο σε πολλά μέρη στην εκλογική μου περιφέρεια όπου η χαμηλή μισθή και ο περίοδος εργασίας οδηγούν σε πραγματική μείωση εισοδήματος για πάρα πολλούς ανθρώπους, οδυνηρές συνέπειες στα μέσα ενημέρωση του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται συνέχεια η τραγική κατάσταση των οικογενειών που πρέπει να καταλήξουν σε τοκογλύφους που έχουν διπλασιάσει τον τζίρο τους μέσα στα τελευταία 4-5 χρόνια και υπάρχει και μια εικόνα της ένδυας και της αθλειότητος. Υπάρχει κάποιος τον οποίο θέλουν να πετάξουν έξω αυτοί που του έχουν δώσει το κατάλληλο στεγαστική ε, ένωση και αν γίνει κάτι τέτοιο τότε τα παιδιά του θα μπουν σε ένα σύστημα περίθαλψης όπου κυριαρχούν οι παιδόφιλοι. Εγώ προσπαθώ να δώσω στους εκλογείς μου ένα εγχειρίδιο για το πώς να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες. Θα ήθελα να ξέρω όμως και εδώ πώς αυτή η τόσο θετική κρίση που θα οδηγούσε στο ενίο νόμισμα και στην τελική οικονομική ένωση Έχετε καταλάβει πώς πλήττει τις οικογένειες στον πραγματικό κόσμο. Πόσο νομίζετε ότι θα χρειαστεί για να υπάρξει μια πλήρης εξέγερση από τους λαούς μας. Η, η Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ. Ε, Έχω πει ότι η οικονομική κρίση επιδίνωσε κοινωνικά προβλήματα. Την περασμένη εβδομάδα είμαστε μια, μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ακούσαμε για αύξηση των αυτοκτονιών, των αμβλώσεων, της ενδοκογενειακής βίας, πάσιμων του κοινωνικού ιστού, ε, πάρα πολλά προβλήματα. Και το ίδιο συμβαίνει και στη δική μου πατρίδα, στην Κύπρο. Και τα ερωτήματα μου είναι πολύ πολύ απλά. Μήπως στο τέλος η Τρόικα και οι δανειστές θέτουν στόχους σε συνθήκες εργαστηρίου ενώ οι κυβερνώντες προσπαθούν να σημειώσουν κάποια πρόοδο ώστε να εξασφαλίσουν την επόμενη δόση με το να γίνονται απολύσεις δημοσίων ή ιδιωτικών υπαλλήλων και εκμετάλλευση εργαζομένων εξορθολογίζονται όντως ε, ο δημόσιος τομέας ε, βλέπουμε πολλέ απολύσει και αυτό έχει αλυσιδωτέ επιπτώσει. Βλέπουμε νέου με πολλά προσόντα να φεύγουν από τι χώρε μα. Και το ερώτημα μου, μιλούμε αόριστα για επανακίνηση τη οικονομίας. Πώς εννοούμε αυτή την επανακίνηση όταν με αυστηρή λιτότητα, με προβλήματα στον τραπεζικό σύστημα, όταν δεν υπάρχουν δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν δεν υπάρχει ένα κλίμα σιγουριάς για να έρθουν επενδυτές και να επενδύσουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα και όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη Πώ μιλούμε ότι θα υπάρχει επανεκκίνηση τη οικονομία, Είναι τραγικά ερωτήματα. Ο κόσμο θα ψηφίσει του χρόνου για τι ευρωεκλογέ και λυπούμε να πω ότι θα στείλουν εκπροσώπους τη χρυσή αυγή, θα στείλουν εκπροσώπους από το κόμμα τη κυρία Μαρή Λεπέν στη Γαλλία και θα ψηφίσουν αυτού που σκέφτονται ευρωσκεπτικιστικά δεν θα ψηφίσουν αυτούς που μιλούν για οικονομική ενοποίηση και για μια καλύτερη και βαθύτερη Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε τραγικά διλήμματα. Ποιε είναι οι λύσεις. Ο Λάγκεν, θέλω να θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, είναι αλήθεια ότι μετά την ε, δημιουργία της χώρας της ζώνης του ευρώ οδήγησε σε πολύ χαμηλότερα επιτόκια για τις χώρες του, του Νότου που δεν χρησιμοποιήθηκαν για μείωση το, της ε, χρέωσης αλλά για αύξηση της κατανάλωσης. Οπότε είναι θέμα ιδίας ευθύνης τους. Δεύτερον, οι μισθολογικές διαφορές. Αν δούμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο παρελθόν είχαν ε, εξασφαλίσει τα συνδικάτα ότι ήταν πολλαπλή η χρήση εργαζομένων στα τρένα από ό,τι χρειάζεται στην πραγματικότητα. Αν δούμε λοιπόν την αυτονομία των συνδικάτων σε ό,τι αφορά τις λογικές ε, διαπραγματεύσεις, μήπως οφείλονται εκεί τα προβλήματα αυτά και όχι στην ευθύνη των κρατών μελών. Και αν θέλουμε να αναφερθούμε στην Ελλάδα, το θετικό στοιχείο της Ελλάδος είναι ο τουρισμός, αλλά δεν μπορεί να έχει κάποιο πλεονέκτημα εναντί χωρών όπως είναι η Κροατία ή η Τουρκία. Επειδή είναι πολύ ακριβή χώρα. Και επίσης, ποια είναι η άποψη κατά τους εμπειρογνώμονες για το τι θα κάνουν τα κράτη. Πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα στην οικονομία, να κάνουν πιο εύκολες επενδύσεις, να κάνουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις και υπάρχει ένα νομικό σύστημα το οποίο είναι σταθερό και μια δημόσια διοίκηση η οποία είναι λειτουργική και υπάρχει έλλειψη διαφθοράς ώστε να πετύχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις ή όχι. Α, μου φάνηκε ότι έχασα τον κατάλογο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το επόμενο πάνελ θα μας εγκαταλείψουν οι διερμηνείς, γι' αυτό θερμή παράκληση σας παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και των δύο πάνελ και υπενθυμίζω ότι το ευρώ υποκατέστησε άλλα νομίσματα και υποθέτω ότι έλαβε υπόσχεση την εμπειρία της διαμορφώσεως και των ισοτιμιών και τις πορείες των άλλων νομισμάτων που επί χρόνια ισχύουν στην παγκόσμια αγορά. Ε, είπαμε με το ευρώ στους Ευρωπαίους πολίτες ότι θα τους εξασφαλίσουμε ένα σταθερό νόμισμα, καλύτερες δυνατότητες δανεισμού και καλύτερη ζωή. Τους είπαμε παράλληλα ότι θα τους εξασφαλίσουμε ορισμένα βασικά ανθρωπίνα δικαιώματα. Ε, δεν ξέρω πόσο επιτύχαμε σε αυτό διότι βλέπω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη περιορίζονται σήμερα σε βαθμό που ε, θα πρέπει να μας προβληματίσει εν ώψη και των ευρωεκλογών που έρχονται και των όσων γίνονται και των όσων διαμορφώνονται πολιτικά μέσα στις κοινωνίες. Έρχομαι να πω για το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τιμπό και πολύ σωστά θα τον παρακαλούσα να ε, μου το αναλύσει αν αυτό οφείλεται ε, στη μείωση των εισαγωγών ή στην αύξηση των εξαγωγών των χωρών του Νότου που θα έχει σημαντική σημασία νομίζω στη συναγωγή συμπερασμάτων και εν προκειμένου να χαιρετήσω και την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου Κάρας να εξετάσουμε τα λάθη τα οποία η Τρόικα έχει κάνει στην διαμόρφωση των ε, πολιτικών ε, στον Ευρωπαϊκό Νότο, διότι τότε θα μας διευθούν και συμπεράσματα, θα, έχουμε σημαντικά συμπεράσματα, τα χρήματα αυτά των δανεισμών των χωρών του Νότου, πού μετακυλήθησαν, πώς διαμορφώθησαν τα ισοζύγια εξωτερικών πληρωμών και αν πήγαν σε άλλες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, χάσαμε ένα κομμάτι από τη μετάφραση. Ευτυχώ επανήλθε και πάλι. Ωραία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να σα ζητήσω να δώσετε σύντομες απαντήσεις. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας διαθέσω πάνω από πέντε λεπτά. Ε, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στο Ζήλο, ο οποίο σεβάστηκε τα χρονικά περιχθώρια που του είχα δοθεί. Ευχαριστώ. Έχουν ε, γίνει πολλέ ερωτήσει και δυστυχώ έχω μόνο πέντε λεπτά στη διάθεσή μου. Δεν θα τι απαντήσω συνεπώ. Ξέρετε, η δική μου άποψη είναι ότι όταν θέσει σε αυτόν σε μία δύσκολη κατάσταση, δεν έχει περιθώρια διαμαρτυρίας αυτού αυτό το έκαναν πολλές χώρες γιατί πριν μπουν σε μια διαδικασία κρίσης είχαν καταγράψει ψηλό εξωτερικό χρέος ε, και αυτό συνέβη σε αρκετές χώρες και όταν είναι πια πολύ αργά ε, ο πόνος είναι πολύ μεγάλος. Τα πάντα τίθονται εκτός ελέγχου σε σχέση με την ε, Ευρωζώνη και προσπαθείτε να χρηματοδοτήσετε επιβάλλοντας φόρους ακόμα και στις επόμενες γενιές. Από την άλλη πλευρά δεν είναι επαρκής η οικονομική ανάπτυξη τότε πραγματικά καλείστε να κάνετε πολύ σκληρές επιλογές. Αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να τονίσω. Αν αποκαλύφθει ότι δεν μπορείτε να πουλήσετε τα προϊόντα σας γιατί είναι πολύ ακριβά, δεν υπάρχει τρόπος να, να τα δώσετε σε χαμηλότερες τιμές. Κανένα, σε κανέναν δεν του αρέσουν οι περικοπές μισθών, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό με οδηγεί σε ένα άλλο σημείο που αφορά την λιτότητα. Βεβαίω συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για τη λιτότητα. Διανύουμε μια περίοδο ύφεση. Εγώ πιστεύω ότι ο πολλαπλασιαστή είναι μεγαλύτερο από το ευρώ. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο υψηλό ε, όσο αυτό που ανέφεραν ορισμένοι. Τι κάνουμε λοιπόν, ξέρουμε ότι βραχυπρόθεσμα η λιτότητα τά καταστρέφει τις θέσεις εργασίας. Συρρυκνώνει στο παρελθόν υπήρχε συμφωνία της Ουάσιγκτον που εφαρμόστηκε από το Δούνου του σε χώρες που είχαν πληγεί από κρίση και η λογική της ε, συμφωνίας της Ουάσιγκτον ήταν η απλή. Δαπανάτε πολλά Συνεπώς θα πρέπει να δαπανίσετε λιγότερα. Ξέρουμε ότι όταν δαπανάτε λιγότερα η ζήτηση θα μειωθεί και αυτό θα καταστρέψει θέσεις εργασίας. Κατά συνέπεια χρειαζόμαστε μια άλλη πηγή ζήτησης για να αντισταθμίσουμε τις απόλυση. Η άλλη πηγή ζήτησης θα πρέπει να, να προέλθει από τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα είναι αντικαθιστώντα τη ζήτηση, ε, την εισαγωγική με ε, ε, χωρία ζήτηση. Πώ το κάνετε αυτό, κάνοντα μία υποτίμηση του νομίσματος. Αυτό Βεβαίως ε, θα εκπλήξω πάρα πολλούς γιατί εμείς ε, οι οικονομολόγοι θεωρούμε θα του ευρώ. Αλλά πιστεύω ότι το ευρώ είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα σε αυτή την κρίση γιατί δεν επιτρέπει τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση να εφαρμόσουν τη συμφωνία της Ουάσιγκτον. Αυτό που κάνετε δηλαδή είναι ότι δεν εφαρμόζεται τη συμφωνία της Ουάσιγκτον εφαρμόζεται την πολιτική που είχαμε στην ε, Γαλλία την εποχή του Ζαν Κλωτρισέ. Όταν ήμασταν στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα η πολιτική αυτή απεκλήθη από τον ΚΡΙΣΕ ε, ο ε, ανταγωνιστικός αποπληθωρισμός. Αντί δηλαδή για να υποτιμήσουμε το νόμισμα υπάρχει μια πολιτική συρρήκνωσης η οποία καλμάρει, καθησυχάζει την οικονομία έτσι ώστε ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από άλλες χώρες. Μάθαμε όμως από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτός ο αποπληθωρισμός χρειάζεται να αυξηθεί πολύ γρήγορα η ανεργία γιατί αυτός ο μηχανισμός αρχίζει να εφαρμόζεται μόνο όταν η ανεργία φτάσει το 20%. Αυτό μάθαμε από αυτές τις χώρες. Ενδεχομένω, άλλες χώρες υπήρξαν περισσότερο τυχερές γιατί είχαν περισσότερο ευέλικτες αγορές. Στις συγκεκριμένε χώρες όμως οι στρατηγικές αποπληθωρισμού ήταν πάρα πολύ δαπανηρές. Ε, αυτό συνεπάγεται το κόστος του να ανοίγει κανεί την Ευρωζώνη. Θα ήθελα τέλος να απαντήσω στα ερωτήματα που ετέθησαν στα γαλλικά από τους ε, συμπατριώτες μου και από τους Βέλγους. Θα απαντήσω λοιπόν στα γαλλικά. Συγγνώμη, μην βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα. Δεν είπα ότι ο πολλαπλασιαστή ήταν μηδέν, ότι υπήρχε ε, ε κατά Ρικάρντο ε, ε, ε, αναλογία, ισοτιμία. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι για να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο χρειάζονται περισσότεροι φόροι, λιγότερε συνεπώς, λιγότερα κίνητρα για εργασία, για επενδύσει, λιγότερη δραστηριότητα. Ε, αναφερόμουν όχι στην αποτελεσματικότητα του κράτους, την οποία αμφισβητώ προσωπικά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου, αλλά αναφερόμουν στις ε, ε, αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Κοιτάξτε, ε, δυστυχώς η οικονομία δεν είναι μια, επιστήμη, μια ακριβής επιστήμη. Θα Μπορούσα όμω να σα παραπέμψω σε άρθρα, για παράδειγμα ένα άρθρο του Ρόκο που υπολογίζει το κόστο ε, τη φορολογία και που δείχνει ότι για ορισμένε κοινωνικο κοινωνικο-οικονομικέ κατηγορίες ε, για παράδειγμα ε, στη Γαλλία βρισκόμαστε στην κορυφή της καμπύλη. είναι τόσο μεγάλη εκτροπή έτσι ώστε αν αυξηθεί αυξηθεί η φορολογία, δεν θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Σε ό,τι αφορά την επίπτωση των ε, ε, ε, μισθών στην ζήτηση εργασία. εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώ δουλειά. Αυτό υπάρχει σε ορισμένες χώρε. Οι κομμουνιστικέ χώρε εγκαθίδρυσαν τη δουλεία γιατί ήταν ο μοναδικό τρόπο για να λειτουργήσουν. Παραπέμπω στο αρχιπέλαγο Γκούλαγκ. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εμπειρία Μισό λεπτό. Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω. Η Ισπανία υπό τον στρατηγό Φράγκο, η μισθή ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Τι παρατηρήσαμε, το ποσοστό ανεργίας ήταν μηδενικό. Η υπήρχε ε, ε, πλεόνασμα μετά το θάνατο του Φράγκο ε, διαπραγματεύτηκαν τα συνδικάτα και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 20%. Δεν υπεραμείνουμε βεβαίως του καθεστώτος του Φράνκο. Δεν πιστεύω ότι το βέλτιστο είναι ένα μηδέν ποσοστό ανεργίας αλλά η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν έχουμε δίκιο να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του κόστου εργασίας και της απασχόλησης. Συγγνώμη, δεν σας διέκοψα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η δουλειά σας. Ο κύριος Τέμπο. Εν συντομία. Αναφέρθηκαν πολύ στην αναθέρμανση της οικονομίας. Νομίζω πρέπει να κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ σκληρή λιτότητα. Με το να καθυστερήσουμε την εφαρμογή αυτής της λιτότητας όμως και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αν είναι καλύτερες οι συνθήκες θα είναι χαμηλότεροι οι πολλαπλασιαστές, τότε μπορούμε να έχουμε καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα με το να καθυστερήσουμε την εφαρμογή της λιτότητας. Το θέμα δεν είναι να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα, το θέμα είναι η διαδικασία λιτότητας να απλωθεί στο χρόνο. Είναι ακριβώς το ίδιο και απαντώ στον Λίαμ που ισχύει και για τους μισθούς. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τους μισθούς. Είναι απλώς να θέσουμε ένα κάτω φράγμα στην μείωση των μισθών. Είναι αρκετά διαφορετικό αυτό από μία αναθέρμανση με την αύξηση των μισθών. Είπα ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο πρότυπο ελαχίστου μισθού στην Ευρώπη και στις χώρες που υπάρχουν πλεονάσματα στο εμπορικό ισοζύγιο να υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις εκεί. Αν δείτε τη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, η Γαλλία δεν έχει κανένα λόγο να αυξήσει τους μισθούς ή τους ελάχιστους μισθούς. Θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει να τους ε, αυξάνει λιγότερο από τον πληθωρισμό ή την ε, παραγωγικότητα, να υπάρξει μια μείωση σε πραγματικούς όρους στη Γαλλία. Αλλά σε χώρες όπως η Γερμανία θα πρέπει να αυξηθούν οι ελάχιστοι μισθοί. Αυτό θα ωφελήσει όλους για να απαντήσω σε αυτά που είπε ο Ζουλ Σαμπόλ. Δεν μπορεί να κάνει κανείς πολύ περισσότερο από το να υπάρξει μια μορφή υποτίμηση σε κάποιες χώρες για να υπάρξει ανάκτηση ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει η αποβιομηχάνηση η οποία κάνει άχρηστες τις προσπάθειες ε, υποτίμηση. εσωτερικής υποτίμησης. Χρειάζεται να έχετε μια βιομηχανία για να έχει κανείς μια ουσιαστική υποτίμηση. Το επιχείρημα όμως δεν είναι ο Ζαν Πολ είναι ο Λαβάλ. Γιατί όταν κάνει κανείς μέσα σε μια συνολική κρίση μείωση των μισθών και γίνεται αυτό από όλους, το τελικό αποτέλεσμα είναι απλώς η μείωση μισθών σε παγκόσμιο επίπεδο. Καταλήγει κανείς σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι γενικά αρνητικό σε όλους και μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεμο. Η Καλή απάντηση λοιπόν στο Λαβάλ είναι η στάση του Κέινς. Όταν θέλουμε να επανεξισορροπήσουμε τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στις χώρες που έχουν ελλείμματα, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να βρείτε και έναν τρόπο να μειώσετε τα πλεονάσματα στις χώρες που έχουν πλεονάσμα. Εάν δεν το κάνετε αυτό, στο τέλος υπάρχει συνολική, συνολικός αποπληθωρισμός και δεν λύνεται το πρόβλημα του ισοσγείου τρεχουσών συνολικών. Πρέπει να δει κανεί όλα αυτά τα πράγματα συνολικά. Η συνένεση τη Washington δεν μπορεί να εφαρμόζεται μηχανιστικά σε όλε τι χώρε και μετά λέμε Α, δεν τα καταφέραμε. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που καταλήγουμε πάντα με αυτό το αδύνατο <clears throat> σχήμα που έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει και ελάχιστο χρόνο απάντηση. Αν θέλουν να στείλουν έγγραφε ε, ε, απαντήσεις οι ομιλητές μας με email ή κάτι τέτοιο θα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι να ακούσουμε τις απόψεις σας. Και επίσης σας ζητήθηκε να δώσετε κάποια άρθρα ή έγγραφα εργασίας ή έγγραφα αναφοράς για τα θέματα αυτά. Έχουμε μόνο ένα τέταρτο καθυστέρηση και θα περάσουμε στο τρίτο πάνελ που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως τα προηγούμενα πάνελ και όπως αυτό που κάναμε πέρσι και πρόπεση για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής υποστήριξης και την επιλεξιμότητα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει πρώτα το λόγο. Ο Σέρβας Ντερούς από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να είστε σύντομοι και οι δύο μιλητές γιατί Έχουμε καθυστερήσει. Αν καταφέρετε να μην ξεπεράσετε τα 7 λεπτά θα σα ήμουν ευγνώμων. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, θα κάνω το παν για να μην ξεπεράσω τα 7 λεπτά. Ίσως μιλήσω υπερβολικά γρήγορα, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθύνω το λόγο στη δική σας Επιτροπή. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτή η συνέβρεση της διαφάνειας και της λογοδοσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάρη στη θέσπιση του ΤΟΥΠΑΚ. Ε, ας μιλήσω για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Τρόικα. Η Τρόικα θα παράσχει βοήθεια σε, επί τη βάση ad hoc. Ρόλος της Κομισιόν στο πρόγραμμα ε, είναι ένας ρόλος που έχει καθοριστεί μέσα από μια διακυβερνητική διαδικασία ε, είναι ένας ρόλος στη διαπραγμάτευση του μνημονίου κατανόησης. Διακόπτη η Πρόεδρος. Όχι, δεν μπορείτε να πείτε τα ίδια με ταχύτερο ρυθμό για να μην ξεπεράσετε τα 7 λεπτά. Πρέπει να επιβραδύνετε και να μην ξεπεράσετε τα 7 λεπτά. Εντάξει, θα το προσπαθήσω, λέει ο κ. Ντερούς. Επομένως, η οικονομική βοήθεια δίδεται από τα χώρες του ευρώ Αυτά έχουν την ιδιοκτησία του προγράμματος αν θέλετε και είναι αυτό βασικό για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Το μοντέλο της Τρόικας έχει αποδειχθεί χρήσιμο, έχει ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συνεχίσουν να ε, συμμετάσχουν στην Τρόικα στο άμεσο μέλλον. Όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος ε, Ρεν, στην ε, συνέντευξη τύπου σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει την ίδια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μελετήσει τη λειτουργία της ε, Τρόικας με στόχο να ενισχύσει την νομοποίηση της Τρόικας και γι' αυτό ως Κομισιόν εμείς παριστάμεθα σε αυτή την ακρόαση, συμμετέχουμε στο διάλογο και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη λογοδοσία. Γι' αυτό το κάνουμε και συμφωνούμε ε, και θα πρέπει να συγχρονιστούμε με τις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Να πω λοιπόν τα βασικά επιτέγματα του προγράμματος. Η επιτυχία είναι αισθητή. Και τελικά το πρόγραμμα έχει αποφύγει την άτακτη χρεοκοπία στις χώρες αυτές έχουν δημιουργηθεί ε, τείχη ασφαλείας που ήταν ε, πολύ σημαντικά. Επιστρέφει σιγά σιγά η ανάπτυξη βάσει των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι περισσότερες χώρες που έχουν κρίση αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις προβλέψεις θα έχουν ανάπτυξη του χρόνου, μισό τα εκατό στην Ελλάδα, μισό της εκατό στην Ισπανία και περισσότερο στην Ιρλανδία και στις άλλες χώρες. Εξαίρεση είναι μόνο η Κύπρος που θα έχει ε, ύφεση 4% το 2014 αλλά θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2015 γιατί τα γεγονότα συνέβησαν αργότερα στη χώρα αυτή. Η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική προσπάθεια που ξεπερνάει το 30% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2009 και για πρώτη πλευρά έχει πλεόνασμα δημοσιονομικό. Στην Πορτογαλία το χρέος έχει μειωθεί στο μισό. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά των ομολόγων και η εμπιστοσύνη έχει σταδιακά αποκατασταθεί. Ε, σιγά σιγά οι χώρες θα μπορέσουν να βγουν οι ίδιες στην αγορά, στις αγορές για να δανείζονται. Αυτό σχεδόν το έχει επιτύχει η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχει διανύσει μεγάλη απόσταση αυτού του δρόμου από το 2015 και μετά εν μέρει η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές, ενώ η Ισπανία την διατήρησε την πρόσβαση στις αγορές όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα βελτιώνεται και η ανταγωνιστικότητα στις χώρες ε, προγράμματος. Το μοναδιαίο εργασιακό κόστος έχει αρχίσει να μειωθεί, ε, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχει περάσει από ε, υψηλό έλλειμμα σε θετικό πρόσημο. Ε, γίνονται μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικές, οι οποίες φέρνουν καρπούς, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ θα μπορούσε να φτάσει στις 6 ποσοστιαίες μονάδες μέσω πρόθεσμα και διπλάσιος μακροπρόθεσμα. Και τέλος, οι τραπεζικοί τομείς έχουν υποστεί ανακεφαλαιοποίηση με μεγάλη πρόοδο κυρίως στην Ιρλανδία και στην Ισπανία και έχει αποφευθεί ε, πιστοτική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, βεβαίως, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ήταν σε γενικές γραμμές ο κατάλληλος παρά τα κάποια σφάλματα και τις κάποιες αδυναμίες του κάθε φορά. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις οικονομικές γιατί είναι ε, κερί μεγάλης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Οι προβλέψεις υπόκειται σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο αναθεώρησης των προβλέψεων αυτών από ό,τι είναι το συνηθισμένο και αυτό δεν θα πρέπει να συγχαίεται με αποτυχία του προγράμματος. Το ότι αναθεωρούνται οι προβλέψεις δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένα ε, το περιεχόμενο του εκάστοτε προγράμματος. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος, Ωστόσο, το βασικό είναι οι εθνικές μεταρρυθμίσεις και οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Έχουμε μια κληρονομιά. Η κρίση αφήνει μια κληρονομιά και αυτό καθυστερεί την ανάπτυξη. Έχουμε απομόχλευση, ε, εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα, ανησυχία, κατακαιρματισμό της αγοράς και αυτό ισχύει κυρίως για τις τράπεζες στα διάφορα κράτη-μέλη οι οποίες δυσκολεύονται να έχουν ε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αν κάνουμε πρόοδο στην Τραπεζική Ένωση, αν έχουμε ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αυτά είναι απαραίτητα πράγματα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομική ολοκλήρωση στη ζώνη του ευρώ. Πρέπει να γίνουν προσαρμογές στους ε, εθνικούς μισθούς. Η πρόοδος ήταν αργή σε κάποιες χώρες και αυτό ε, δεν οδήγησε τελικά σε πτώση των τιμών στην αγορά. Έχει αυξηθεί η ανεργία και υπάρχει ακαμψία στις αγορές προϊόντων που απαιτούν περισσότερο ανταγωνισμό και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όντω, η κατάσταση στο επίπεδο τη απασχόληση παρουσιάζει πάρα πολλέ προκλήσει και αυτό το γνωρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλαβε δράση για να καταπολεμήσει αυτό το τεράστιο ποσοστό ανεργία των νέων. Έχουμε το σύστημα εγγυήσεων που προσφέρεται στου νέου. Ε, σταθεροποιείται ε, αυτό αυτή, αυτό το ποσοστό ανεργίας των νέων στις περισσότερες χώρες και δεν αυξάνει δραματικά πλέον, έχει σταθεροποιηθεί κάπως. Είναι σημαντικό το, ότι οι προσερμογές που είναι αναπόφευκτο να γίνουν να μοιραστούν ισότιμα με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο ε, τρόπο και η επιλεξιμότητα, η αιρεσιμότητα ε, πάντοτε έχει ως στόχο να ε, μην επιβαρύνει τους, τις περισσότερο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να προστατευτούν οι πιο ευπαθείς οι κερδοφόρες επιχειρήσεις ε, και η μεγάλη ακίνητη περιουσία έχουν ε, υπόκεινται σε φορολόγηση και έχουν αυξηθεί αντίστοιχοι συντελεστές έτσι ώστε όλοι να επομιστούν το βάρος που τους αναλογεί. Είναι δύσκολα αυτά τα μέτρα, αναπόφευκτα όμως οι χώρες είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόντουσαν πριν από τρία χρόνια και αποφεύθηκε η ε, αποφεύθηκαν οι άτακτες προσαρμογές οι οποίες θα ήταν πολύ πιο επίπονες για τον Ευρωπαίο πολίτη. Θεωρώ ότι, θεωρούμε ότι σταθεροποιείται η κατάσταση και ήδη λίγαν συντόμως θα υπάρξει έξοδος από μνημόνιο για Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. Η κρίση του εθνικού χρέους είναι ε, σημαντική. Ε, εάν έχουμε τραπεζική ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό θα είναι θεμελιώδες για να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη στο σύστημα και να ενισχυθεί, να πυροδοτηθεί εκ νέου η οικονομική ε, δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ. Γλιτώσαμε κανένα λεπτό. Ο Κλάους ε, Μαζόχ από την Οικονομική Υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι. Μπορεί, μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο σας ή ο προηγούμενος. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Μπορώ να συμφωνήσω με τη δήλωση της Κομισιόν του κ. Ντελός, ιδίως για τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την ε, κοινωνικά ισοδίκαια μορφή των προγραμμάτων αυτών. να σας αναφέρω τις απόψεις μου σε σχέση με την πρόοδο που επιτεύχθη στις χώρες κρίσης με το πρόγραμμα αυτό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ισπανίας. Εγώ φυσικά βασίζομαι στη δική μου εμπειρία στην ανάλυση των ε, εξελίξεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με την Κομισιόν δίδουν τεχνική αρρωγή προσφέρουν συμβουλές στην Ευρωομάδα και στις εθνικές κυβερνήσεις. Αλλά είναι το Eurogroup το σώμα το οποίο παίρνει τις αποφάσεις για το πώς θα δοθεί χρηματοδοτική βοήθεια, κατά από ποιους όρους και πώς. Ήταν υψηλό το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της κρίσης και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού των χωρών κρίσης έχουν αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το κόστος ήταν αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και κυρίως το κοινωνικό κόστος ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων οικονομικών ανισομεριών και των διαρθωτικών ακαμψιών που τους επιτράπει να συσσωρευτούν στις χώρες αυτές πριν από τα προγράμματα προσαρμογής από το 2008 και επέκεινα. Κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία είχε υπερβολική άνοδο του ιδιωτικού του του ιδιωτικού της χρέους και δημιούργησε μεγάλα ε, ελλείμματα χωρίς να επιτύχει τους στόχους τους. Άλλες χώρες όπως η Ελλάδα είχαν μεγάλες αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες ιδίως σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις από την ε, είσοδο στο ευρώ έχουν φτάσει σε, έφτασαν σε πολύ ψηλό δημόσιο χρέο, το οποίο δεν ήταν ιδιώσιμο. Αυτό οδήγησε σε υπερθέρμανση τη οικονομία και απώλεια ανταγωνιστικότητα. Ενώ συγχρόνω υπήρξαν σημαντικέ ε, ακαμψίε, ιδίω προ τα κάτω των μισθών και των ε, τιμών που δεν εμπόδισαν την εύκολη εφαρμογή της προσαρμογής και οδήγησαν σε αύξηση της ανεργίας. Σε άλλες χώρες όπως ήταν η Ιρλανδία, η η φούσκα στις αγορές, ε, στη στεγαστική αγορά υπονόμευσε την βιωσιμότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οδήγησε σε τεράστιο χρέος των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αλλάζουν οι πηγές της κρίσης σε πολλές χώρες, αλλά παντού υπήρξαν μεγάλες ανισομέρειες και ακαμψίες που έπρεπε να διορθωθούν για να μπορέσει να υπάρξει βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν υπήρχε καμία εναλλακτική λύση στη δημοσιονομική εξυγίανση, στην απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και τις διαφορετικές αλλαγές για να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα. Υπήρξαν φυσικά και ε, δυσκολίες στο να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές οι οποίες αύξησαν και το κόστος. Η καθυστέρηση αυτή και η μη σωστή εφαρμογή μετά από την εφαρμογή των προγραμμάτων, ιδίω στην Ελλάδα, ήταν και αποτέλεσμα μιας ε, ε πολιτικής ε, στάσης από ορισμένους τομείς που δεν ήθελε να υποστηρίξει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Όλες οι χώρες όμως μέσα σε αυτά τα προγράμματα έχουν πετύχει σημαντική πρόοδο στο να μειώσουν τις οικονομικές τους ανισομέρειες και να αντιμετωπίσουν τις ακαμψίες και να εξασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική ισορροπία. Έχουμε λοιπόν μια βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον. Μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η πρόοδος δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς, τα προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας. Όπως ελέγχθη λοιπόν και προηγουμένως, η κατάσταση <clears throat> μεταξύ 2009 και 2013 είχε σημαντικά ε, επιτέγματα. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα έχει βελτιωθεί στην Ελλάδα κατά 12% και κατά 6 με 8% στις άλλες χώρες, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Είναι μικρότερη η πρόοδος στην ε, Κύπρο γιατί μόλις πρόσφατα ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό. <clears throat> Η προβλέψη είναι ότι η Πορτογαλία και η Ιρλανδία θα έχουν πρωτογενές πλεόνασμα το 2014 ενώ η Ελλάδα θα μπορέσει να έχει ένα τέτοιο πλεόνασμα ήδη εφέτος. Όλες οι χώρες του, των προγραμμάτων αυτών για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους στην Ιρλανδία. Το μοναδιαίο εργασιακό κόστος από το 2008 σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 20%. Είναι πολύ θετικά επίση τα στοιχεία ανταγωνιστικότητα, διότι ήταν χαμηλός ο πληθωρισμός στι χώρε αυτέ, ακόμα και αρνητικός στην περίπτωση της Ελλάδος από την άνοιξη του 2013 όπως αναφέρθηκε και από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αντιμετωπιστήκαν οι αντισωμέρειες στο ισοζύγιο τρέχουσων πληρωμών, οι οποίες ήταν αξιοσημείωτες τις προσπάθειες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ανακεφαλαιωθεί και αναδιαρθωθεί. Είναι στη διαδικασία αυτή και έχουν επιτύχει χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και η οικονομική ανάπτυξη στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία θα γίνει θετική εφέτος. Στην Ελλάδα η οικονομική ανάπτυξη ελπίζουμε ότι θα επανέλθει στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Γενικά τα προγράμματα αυτά έχουν λειτουργήσει θετικά, έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες βάσεις για μελλοντική δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη, παραμένουν όμως προκλήσεις. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να, να συνεχιστεί, να υπάρξουν αποθέματα στο δημόσιο προπολογισμό ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κοινωνικό κόστος των περαιτέρω των μελλοντικών οικονομικών κλειδονισμών δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο σε αυτή την κρίση πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσει και για την αγορά για να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και χαμηλότερες τιμές για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών και επίσης να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και των καταναλωτών. χωρί αυτέ τι μεταρρυθμίσεις στις αγορέ προϊόντων η πραγματική μισθή και η απασχόληση θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο για πάρα πολύ καιρό διάστημα. Χρειάζεται μια πιο προορατική λοιπόν αντιμετώπιση από τι εθνικέ κυβερνήσει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και τη διαφθορά και μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο για να αντιμετωπίσουμε μια μεγαλύτερη και να έχουμε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και μεγαλύτερη κοινωνική ισοδικία. Υπάρχει ένα κίνδυνο να γίνει διαθωτική η τωρινή ε, ανεργία και να υπάρξει διάβρωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους νέους. Υπάρχει οδητός χαρακτήρας των αγορών εργασίας και θα πρέπει να περάσουν οι ανθρώπινοι πόροι από μη εμπορεύσιμες σε εμπορεύσιμες ε, εργασίες και υπηρεσίες και να γίνει πιο εύκαμπτη η οικονομία των χωρών αυτών. Επίσης, οι χώρες αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των τραπεζών του ώστε να μπορέσουν οι τράπεζε αυτές να διευκολύνουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε πιστώσει της πραγματικής οικονομίας, ιδίως στις μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Οι απαραίτητε λοιπόν ενέργειες θα πρέπει να κινηθούν προς το να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση ρευστότητα κεφαλαιοκική επάρκεια των τραπεζών και μεγαλύτερη κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης όλε αυτέ οι προκλήσει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη ταχύτητα και με αποφασιστικό τρόπο γιατί παρά το γεγονό ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κόπωση σε σχέση με τι μεταρρυθμίσει, θα πρέπει να εδραιωθούν τα επιτευχθέντα και να προχωρήσουμε με την υπόλοιπη ατζέντα μεταρρυθμίσεω στι χώρε αυτέ. Το να καθυστερήσουμε αυτέ τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει δεν θα ωφελήσει, θα θέσει σε κίνδυνο όλο το πρόγραμμα αυτό και δεν θα δημιουργήσει τι βάσει για ανάκαμψη τη απασχόληση και τη οικονομία στι χώρε αυτέ. Και μετά στη διάθεσή σα για ερωτήματα, εάν έχετε πια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε έναν κατάλογο από άτομα που θα ήθελαν να διατυπώσουν ερωτήσεις. Νομίζω ότι δεν, δεν είναι σκόπιμο να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις. Ας ε, τις βάλουμε λοιπόν σε ομάδες σε τριών ή τεσσάρων ερωτήσεις. Έχουμε λοιπόν τους τρεις πρώτους ε, ομιλητές. Ο τρίτος είναι ο κύριος Στυλακάκης ε, θα δώσουμε το λόγο για απαντήσεις και θα προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε κάπως το χρόνο μας. Θερμή παράκληση, όχι παραπάνω από 1,5 λεπτό η ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι άκουσα αυτά που είπε όλη η Ρεν σήμερα το πρωί σε σχέση με την αξιολόγηση της ε, Τρόικας, κάτι το οποίο το χαιρετίζω εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι επίσης αυτή η ακρόαση θα πρέπει να αφιερωθεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Τρόικα δεν λειτουργεί με ένα διαφανή τρόπο, δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση, δεν έχει δημοκρατικό έλεγχο και είναι ένα διακυβερνητικό εργαλείο και όχι ένα ενωσιακό εργαλείο. Θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο ρόλος των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στην Τρόικα ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ τους και ποιες είναι οι σχέσεις τους με τα κράτη-μέλη τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία της Τρόικας. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία κάνει η Τρόικα, πώς δίνει αναφορές, πώς ε, γίνεται η πραγματοποίηση των μέτρων που προτείνει η Τρόικα, πώς ακολουθεί τι διαδικασία ακολουθούν οι επαφές των κρατών μελών με την Τρόικα. Ποιο είναι το έδαφος επί του οποίου εδράζονται οι προτάσεις της Τρόικας και οι αποφάσεις της Τρόικας. Και πώς βλέπει η Τρόικα τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη τα οποία εμπλέκονται στα προγράμματα αυτά. Και το τελευταίο μου ερώτημα, πώς αντιμετωπίζει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας εικόνας που υπάρχει για την Τρόικα και της δικής τους εμπιστοσύνης και ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν για την συνέχιση της εργασίας τους και τη συνεργασία με την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Όλοι Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή και την Κεντρική Τράπεζα γιατί η πολιτική σας έχει ένα πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που θυμίζει λίγο ανακριτική επιτροπή. Ποιες είναι, σε τι, ποια βάση χρησιμοποιήσατε για να αποφασίσετε τα μέτρα που υιοθετήσατε, καταρχάς ποια είναι η αξία του πολλαπλασιαστή. Μιλήσατε πριν από λίγο για διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ποια είναι αυτή η ελαστικότητα που διατηρήσατε για να μπορέσετε να εφαρμόσετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ερώτημα προς την ΕΚΤ. Έχετε σχεδόν την πλειοψηφία του ελληνικού χρέους. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιο μέρος ε, χρησιμεύσε από, τα, ε, από το χρέος για να ε, εξυπηρετήσει. Ε, γνωρίζουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα δίνει ένα μέρος ε, για να βελτιώσει τον προπολογισμό της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Τέλος, είναι ρόλος Κεντρικής Τράπεζα σε αυτό το πλαίσιο να δίνει συστάσεις πολιτικής του προπολογισμού και φορολογικής πολιτικής. Θα ήθελα να πω ότι με λυπή η απουσία του Δούνου του υπάρχουν σορισμένα στοιχεία που θα θέλαμε να διευκρινίσουμε. Μία ερώτημα και για τους δύο. Πιστεύετε ότι με την εφαρμογή του ΕΜΕΣ υπάρχει ένα έμβριο για το μέλλον και η, ε, Thank ε, είναι Ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Θα μιλήσω λοιπόν για ένα συγκεκριμένο θέμα. Μιλήσατε για την ελληνική περίπτωση, για την αντίσταση στις αλλαγές και συμφωνώ μαζί σας. Το ερώτημα μου είναι πώς εσείς αντισταθήκατε σε αυτή την αντίσταση στις αλλαγές. Γιατί τα τελευταία αυτά χρόνια χρηματοδοτήσατε τον ελληνικό δημόσιο τομέα και καταστρέψατε τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι το ουσιαστικό μου ερώτημα. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα δεν έδωσε σχεδόν τίποτα για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Όλοι τους προήλθαν από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που συνέβη στον ιδιωτικό τομέα είναι ότι συνδεξιδοτήθηκαν ε, πρόωρα, ενδεχομένως ε, μερικοί γύρω στα 50. Η Επιτροπή δεν θέλει καν να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Πόσοι άφησαν τον ε, δημόσιο τομέα. Βεβαίω λέτε ότι υπήρχε αντίσταση, αλλά αυτή χρηματοδοτήθηκε με δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα στραγγαλίστηκε ο ιδιωτικός τομέας που δεν έχει ρευστότητα. Όλη η ρευστότητα διοχετεύεται σήμερα στο δημόσιο. Το ερώτημά μου συνεπώς είναι για ποιο λόγο το κάνατε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θα πρότεινα να κάνω τώρα είναι να δώσω στους ομιλητές τέσσερα λεπτά για να μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα και μετά να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Ποιος θα ήθελε να πάρει πρώτο το λόγο. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που μου ετέθεσαν. Θα απαντήσω για την ε, λογοδοσία της ε, Τρόικα και για την ε, Τρόικα. Θα μπορούσε να απαντήσει και ο συνάδελφός μου. τώρα, λογοδοσία της Τρόικας. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου. Όπως είπα, η Τρόικα δημιουργήθηκε από τις χώρες μέλη για ειδικού σκοπούς και λόγω κάποιας ανάγκης, για να το πούμε το όνομά του. Το σύστημα της Τρόικα προσαρμόστηκε και ενεκρίθη το Μάιο του 2013 και αυτό επιβεβαίωσε ότι όταν βοηθούν με τις χώρες θα πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του ε, ε, Δουνουτού και της ΕΚΤΕ. Μολονότι εκείνη την εποχή δεν υπήρξε κάποια πρόβλεψη, σιγά σιγά οι νομοθέτες το πρόβλεψαν και υπάρχει τώρα μια νομική βάση για τις δραστηριότητες στην Τρόικα. Σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία είναι σαφές ότι το κάθε θεσμικό όργανο έχει ένα διαφορετικό είδος λογοδοσίας και διαφορετικούς ε, συμφεροντούχους. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, ε, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ε, λογοδοσία περνάει από τον Αντιπρόεδρο στο Κοινοβούλιο και ο Αντιπρόεδρος σας επισκέφτηκε εδώ σε πολλές ευκαιρίες να συζητήσει τα προγράμματα την περίπτωση της Κύπρου που ήρθε στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσει το πρόγραμμα και βεβαίως είναι έτοιμος να επανέλθει στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή σας ή στην Ολομέλεια για να μπορέσει να εξηγήσει την απόφαση της Επιτροπής από κοινού με τις χώρες μέλη. Να δώσει δηλαδή συγκεκριμένες εξηγήσει και με αυτόν τον τρόπο να τεθεί το θέμα της λογοδοσίας. Φαντάζομαι ότι τα πιο σημαντικά θέματα θα πρέπει να συζητηθούν αργότερα στα πλαίσια της ίδιας πρωτοβουλίας. Το θέμα για τους πολλαπλασιαστές. Κάθε... Αυτό είναι ένα θέμα που συζητήθηκε εκτενώς στο παρελθόν. Η Επιτροπή αναγνώρισε νωρίς ε, ότι οι πολλαπλασιαστές σε περιόδους κρίσης είναι υψηλότεροι από ό,τι υπό φυσιολογικές συνθήκες. Βεβαίως είναι ιδιαίτερα τεχνικό αυτό το θέμα, αλλά όταν η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε σημείο μηδέν, εάν υπάρχουν περιορισμοί εσωτερικοί, αν η οικονομία είναι αποδυναμωμένη, τότε ε, είναι υψηλότεροι οι πολλαπλασιαστές από ό,τι συνηθίζεται. Γνωρίζουμε και υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των τριών ότι οι πολλαπλασιαστές είναι διαφορετικοί ανάλογα με το ε, τύπο των μέτρων που υιοθετούνται. Ξέρουμε ότι τα μέτρα ε, ε, για τις δαπάνες έχουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές. Από την άλλη πλευρά είμαστε υπέρα γιατί είναι μια πιο διαρκής προσαρμογή. Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι όλες οι μακροοικονομικές προβολές που βρίσκονται στη βάση του των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της μεταρρύψης συζητώνται με τις χώρες μέλη και βασίζονται σε μια κοινή σειρά από προβολές και σε μια κοινή σειρά πολλαπλασιαστέ. Χρησιμοποιούμε συνεπώ στις χώρες ακριβώς του ίδιου ε, πολλαπλασιαστέ με τους συναδέλφους από, το, από την άποψη λοιπόν αυτή έχουμε την ίδια προσέγγιση. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στο τελευταίο ερώτημα γιατί ο χρόνος πιέζει που αφορά το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Αυτό που κάναμε είναι πρωτίστως εστιασμένο στην ε, εξυγίαση στην Ελλάδα λαμβάνοντας ε, υπόψη την υπερχρέωση στην ε, χώρα αυτή. Μία από τις βασικές προτεραιότητες ήταν η εξυγίαση και η βιωσιμότητα του κρέους. Αυτή ήταν η βασική προτεραιότητα και το λόγο αυτό επενεργήσαμε ιδιαίτερα στις, στον, του, στον τομέα των συντάξεων και των μισθών. Ε, συνεπώς είναι φυσικό τα δύο αυτά στοιχεία να είναι τα πιο ε, σημαντικά σε ό,τι αφορά τη ρύθμισή τους. Ε, ασχοληθήκαμε λοιπόν με, τον, το δημόσιο. Η, το μνημόνιο από κοινού με τις ελληνικές αρχές προβλέφθηκαν και άλλα ε, μέτρα, ε, η εθελουσία έξοδος ε, για παράδειγμα, η αναλογία μεταξύ των συνταξιοδοτούμενων και των προσλήψεων. Νομίζω ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε πρόσφατα. Συνεχίζονται παρόλα αυτά οι συζητήσεις σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα στο δημόσιο δεν έχουμε εγκαταλείψει το δημόσιο. Εμεί θέλουμε να μετακυλήσουμε πόρους από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Ο, δημόσιο δημόσιος τομέας ήταν υπερδιωγωμένο. Uh, ο κύριο Μαζούχ παρακαλώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον Σερβάς Ντερούς και θα ήθελα να προσθέσω κάτι για τον δημόσιο τομέα. Πρώτα είχαμε πολύ μεγάλες μειώσεις μισθών και συντάξεων δημοσίου και όπως είπε και ο Σορβάς, οι μειώσεις αυτές ήταν προοδευτικές, δηλαδή ήταν μεγαλύτερες για τους υψηλόμεσθους παρά για τους χαμηλόμεσθους. Επομένως και ο δημόσιος τομέας επλήγει, χρειάστηκε να υποφέρει αυτές τις, όλες αυτές τις, ε, τη δημοσιονομική προσαρμογή τώρα για τις απολύσεις. Πράγματι, δεν έχουν προχωρήσει με τόσο γρήγορο ρυθμό και δεν ήταν τόσο επιτυχημένη η πρόοδος όσο είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση στον τομέα αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, βρίσκεται εν εξελίξη. Υπάρχει νέος υπουργός ε, διοικητικής μεταρρύθμισης. Ο κύριος Μητσοτάκη, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολο το έργο του. Έχει δρομολογήσει αυτή τη διαδικασία και έχει αναλάβει δέσμευση για περισσότερο streamlining, για περισσότερη ευθυγράμμιση και για μείωση του όγκου του δημοσίου τομέα. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα του πρώτου ομιλητή και του δευτέρου. Ε, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα. Και μπορώ να σας πω το εξής. Ο Σερβάς σας περιέγραψε τη διαδικασία. Βάσει της συνθήκης η Κομισιόν είναι το liaison, η σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπολείπων για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Και όπως ε, ανέφερε και ο κύριος Μάριο Ντράγκη, είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μέρος της Τρόικας σε καιρούς τόσο ε, χαλεπούς κρίσης. Δεν παρέχουμε χρηματοδότηση ούτε οικονομική βοήθεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για χώρες όπως η Ελλάδα κυρίως, αλλά και η Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, έχουμε ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, στηρίξει ε, τη ρευστότητα του τραπεζικού τομέα, άρα έχουμε παράσχει οικονομική στήριξη ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδιαιτέρως να είναι μέρος της Τρόικα, διότι μπορούμε να συμβάλλουμε με την εμπειρογνωμοσύνη μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο μηχανισμός ε, μεταφοράς της νομισματικής πολιτικής είναι στρεβλός στη ζώνη του ευρώ. Είναι κατακαιρματισμένος ο χρηματοπιστωτικός τομέας και άρα είναι δύσκολο ε, οι αλλαγές νομισματικές, ε, νομισματικής πολιτικής που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ να φτάσουν με ισότιμο τρόπο σε όλες τις γωνιές της ζώνης του ευρώ συζητούμε με τις εθνικές αρχές, συζητούμε με το Eurogroup, χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είναι πολύ σημαντικές και είναι και μια πολύ θετική παρενέργεια θα έλεγα, γιατί θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ευελιξία και γιατί οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματα στην μετάδοση ε, των ε, ε, αποφάσεων της νομισματικής πολιτικής. Έχουμε ανακεφαλαίωση του τραπεζικού τομέα με τη βοήθεια των προγραμμάτων στις χώρες αυτές και πολλά προβλήματα που υπάρχουν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Έχει μειωθεί η δυσχερή θέση. Τα οικονομικά προβλήματα είναι λιγότερο ε, ε, οξέα για τις χώρες αυτές από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εγώ. Τα μέλη μπορούν να ξαναπάρουν το λόγο στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Κέρτ Γιάν, Εμπίν Φίλιπ Λαμπέρτς, Μαρίσα Ματέ, Έλα, είναι οι επόμενοι ε, βουλευτές που θα θέσουν ερωτήματα. Παρακαλώ. Όταν ακούω τους δύο ομιλητές που είναι καλεσμένοι μας, είναι σαν να μιλάει κάποιο εκπρόσωπο τη Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, να δούμε ποιε είναι οι υποθέσει επί των οποίων βασίζονται οι προβλέψει του που έχουν διαψευστεί οι περισσότερε. Λέγανε ότι η Ελλάδα θα είχε αύξηση 1,1% το 2012 όταν υπήρξε ύφεση 6,4, τεράστια διαφορά. Το, 2011 λέγανε μείον 2,6 ενώ στην πραγματικότητα ήταν 7. Για την Ελλάδα επίσης έλεγε ότι θα αυξηθεί στα 245% και 250% το 2012, αλλά τώρα μετά, αν συμπελάβουμε την αναθίαρθρωση, είναι 169%. Το ίδιο φαινόμενο ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της, του Μεσογείου. Λοιπόν, οι προβλέψεις σας είναι χειρότερες από τις προβλέψεις καιρού που έχω από τις χειρότερες προβλέψεις καιρού που έχω ακούσει. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα καχύποπτος για οικονομολόγους που έρχονται από συγκεκριμένους φορείς. Λέτε ότι είναι επιτυχία ο χαμηλός πληθωρισμός, ενώ πάμε προς αποπληθωρισμό και όλοι έχουν κρούσει το, το κόδωνα του κινδύνου ότι κινδυνεύουμε να πέσουμε στη λούμπα της Ιαπωνίας. Γιατί λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, γιατί έχετε υποτιμήσει τη φύση της κρίσης, είσαστε οικονομολόγοι, έχετε σπουδάσει σε καλά πανεπιστήμια, δουλεύετε για σοβαρούς φορείς. Μήπως ήταν ε, κατά κάποιο τρόπο ευσεβείς πόθη αυτά τα οποία σας οδήγησαν στα συμπεράσματά σας. Όταν θεωρείτε ότι το ευρώ είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα προσπαθήσατε να πείσετε το κοινό στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι τώρα έρχεται, αυτή τη στιγμή τώρα θα έρθει η ευμάρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι τα λαθασμένα στοιχεία οδήγησαν σε λαθασμένη αξιολόγηση, σε λαθασμένες προβλέψεις, σε λαθασμένες προσδικίες, σε λαθασμένη θεραπεία που έχει σπρώξει τις χώρες από την οικονομική τελμάτωση στην κρίση, την πολιτική κρίση που δεν τους επιτρέπει πια να κάνουν διαρθρωτικές αλλαγές. Οι νέοι αυτών των χωρών βασανίζονται πια από την ανεργία και είναι στο κατόφλι της κοινωνικής έκρηξης. Εγώ δεν βλέπω έξοδο από το τούνελ όπως βλέπετε εσείς με τις λανθασμένες σας προβλέψεις. Δυστυχώς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη φορά που ξεπεράσατε το χρόνο σας γι' αυτό σας άφησα. Αλλά μην το πάρετε για προηγούμενο. Μην το ξανακάνετε. Ο Φιλίπ. Σας ευχαριστώ. Ε, γιατί είπατε πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα εγώ ορισμένα πράγματα. Μας λένε δύο ομιλητέ μας ότι κατά κάποιο τρόπο κάνουμε λάθος ακρόαση. Δεν είσαστε οι λήπτες αποφάσεων, εσείς δίδετε κάποιες ε, προτάσεις στην Κομισιόν και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις είναι το Eurogroup και εξάλλου γιατί κάνουμε μια ακρόαση αφού όπως λέτε θα επανέλθει η ανάκαμψη. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Συγκεκριμένα ερωτήματα τώρα. Λέτε ότι είσαστε απλώς τεχνοκράτες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιστεύει ότι οι επιστολές του Ντράγκη προς την Ιταλία, προς την Ιρλανδία, προς την Πορτογαλία είναι καθαρά τεχνοκρατικές συμβουλές ή ήταν κάτι περισσότερο. Για μένα ήταν περισσότερο πολιτική περιορισμή, δεν ήταν τεχνική τεχνικές συμβουλές. Μπορεί να ασφάλω και για τους δύο σας. Ποιο δίνει τι εντολές. Και αυτό είναι το ερώτημα του Όθμαρ Καράς που δεν το απαντήσατε. Ποια είναι η εντολή σα. Γιατί αυτά που είπε ο προηγούμενο ηγέτη του Eurogroup. Είπατε ότι δεν του δίνουμε καμιά εντολή και υπάρχει απλώ ένα μνημόνιο κατανόηση. Λοιπόν, εσεί αποφασίζετε και τα δέχετε αυτά που κάνετε το Eurogroup ή όχι. Πέστε μα. Η ανάλυση βιωσιμότητος του χρέους. Κύριε Σερβάστερός, μας είπατε ότι τελικά αυτή η ανάλυση είναι τελικά θέμα πολιτικής εκτίμησης όταν ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σας υποχρέωσε την διεύθυνση της Κομισιόν να δεχτείτε την φανταστική αυτή ιδέα ότι το 2010 θα μπορούσε να είναι το ελληνικό χρέος. Η Κεντρική Τράπεζα ήθελε να το κάνει αυτό και εσείς τελικά δεχτήκατε την άποψη αυτή τη Κεντρική Τράπεζα ω Κομισιόν. Μπορείτε να μα πείτε κάτι περισσότερο για όλα αυτά. Και το τελευταίο ερώτημα, <clears throat> και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο προλαλή σα. Κάνετε κάποιε προβλέψει, αλλά λαμβάνετε υπόψη το μη γραμμικό χαρακτήρα που μπορεί να προκύψει λόγω μια έκρηξη στι χώρε αυτέ ή θεωρείτε ότι τα πράγματα λειτουργούν όπω λένε οι προβλέψει σα. ζητώ Παρακαλέσαν να περιοριστείτε σε 1,5 λεπτό. Η Μαρίζα, είναι πολύ καλό που έχω την ευκαιρία να, θέσω ερωτήσει στην Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κρίμα που δεν είναι εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το θέμα που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η λογοδοσία σε δημοκρατικό επίπεδο. βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τρόικα δεν εμπλέκει καθόλου τους πολίτες των χωρών που, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη σε σχέση με το επίπεδο επίτευξη στόχων από τις χώρες αυτές που βρίσκονται στα μνημόνια. Γιατί υπήρξε ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα στις χώρες αυτές, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν είναι μονάχα η λιτότητα η οποία έχει ε, αποτύχει, αλλά ότι έτσι κι αλλιώς το σύνολο των ε, πολιτικών σας είναι λαθασμένες. Έχετε κάποιους δικούς σας δείκτες, αλλά οι δικοί μας δείκτες δείχνουν κατάφορα μία ε, ύφεση, ένα τεράστιο αριθμό ανέργων, ατόμων που μεταναστεύουν από τις χώρες μας για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται. Υπάρχει μια καταστροφή η οποία, την οποία υπέστησαν οι χώρες αυτές χωρίς να υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Εσείς είσαστε χειρότεροι και από τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Είναι πολύ πιο προβλέψιμος ο καιρός από αυτό το οποίο έχετε κάνει εσείς. Ο κύριο Δερούς είπε με σαφήνεια ότι το πρόγραμμα της ε, της ε, Τρόικας είναι <clears throat> μια λύση, αλλά τελικά αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεστε την κρίση για να μετακυλήσετε τους πόρους από τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και στις τράπεζες κτλ. Και θα ήθελα κλείσω εδώ κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα αποδεχτείτε για πάντα ότι το πρόγραμμα της Τρόικας δεν έχει πετύχει κανένα στόχο οικονομικό, αλλά απλώς είναι μια διαδικασία ιδεολογικής προσαρμογής στις χώρες του Νότου. Αγαπητοί συνάδελφοι, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Σας παρακαλώ να βρείτε υπόψη σας ότι περιορίζεται και ο χρόνος που έχουν οι φιλοξενούμενοι μας για να απαντήσουν. Είναι, η κυρία Τζαβέλα. Κυρία Τζαβέλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο κυρίους για την παρουσία τους και την ενημέρωση που μας κάνουν. Ε, ε παρατηρώντας ε, χώρες που είναι σε μνημόνιο ε, βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι κάθε μία από τις χώρες αυτές λίγο πολύ έχει ακολουθήσει ένα πρόγραμμα το οποίο υπέδειξε η Τρόικα. Παρά το γεγονός αυτό, δηλαδή μείωση μισθών, μείωση εργοδοτικών ε, εισφορών, ε, θέμα ε, φοροδιαφυγής, ε, μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν αν δούμε προσεκτικά όλες τις χώρες αυτές δεν έχουν προσελκύσει μέχρι τώρα μία σοβαρή μεγάλη επένδυση. Καμία. Ακόμα και αυτές οι οποίες πάνε καλά. Και η ερώτησή μου είναι γιατί. Και δεν είναι μόνο το διεθνές κεφάλαιο που δεν ελκύεται προς αυτές τις χώρες παρά το γεγονός ότι έχουν μειωμένο εργασιακό κόστος ούτε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια δεν κατευθύνονται για επενδύσεις στις χώρες αυτές. Για ποιο λόγο λοιπόν. Ωραία. Θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις. Πολλές από τις ερωτήσεις συμπίπτουν. Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ στα μέλη για τις ερωτήσεις που απίφθηναν. Θα απαντήσω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα όλες τις ερωτήσεις. Καταρχάς σε ό,τι αφορά το θέμα των προβλέψεων. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα εδώ. καταλαβώ τον προβληματισμό σε ό,τι αφορά την ποιότητα των ε, προβλέψεων που αφορούν το πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα θέμα που λαμβάνει υπόψη τη σοβαρά η Επιτροπή. Ε, τα, οι προβλέψεις ε, είναι η βάση για την οικονομική εποπτεία και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είναι όσο γίνεται πιο καλή η πρόβλεψη. πρόβλεψη. Ενδεχομένως μπορεί να αποτύχουμε, κανένας δεν είναι τέλειος. Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές προβήκαμε σε πάρα πολλές αναλύσεις ό,τι αφορά την ακρίβεια των προβλέψεων και θα πρέπει να πω ότι οι προβλέψεις επιτροπής έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο ακρίβειας. Αυτό μια γενική αρχή. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες χώρες, είπα από την αρχή ότι στις χώρες αυτές σε σε κρίσης και αβεβαιότητας το ενιαίο νόμισμα, οικονομική όταν δεν, όπου δεν υπάρχουν μηχανισμοί διακυβέρνησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν οποιασδήποτε προβλέψεις. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την κατανοησή σας και όχι την κριτική σας θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι προβλέψεις αυτές γίνονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Αυτό το βλέπουμε και για τις χώρες αυτές. Οι προβλέψεις συμφωνίας δεν ήταν καλύτερες από τις δικές μας. Να επανέλθω στην Ελλάδα. Ε, δεν, τα, ε, δεν στοχεύσαμε, αλλά για άλλους λόγους. Για τις ευάλωτες χώρες υπάρχουν πολλά καινούρια στοιχεία. Έχουμε ε, θέματα που αφορούν το κράτος και το τραπεζικό τομέα. Έχουμε μετακινήσεις ε, του οικονομικού κινδύνου. Έχουμε ε, φαινόμενα μετάδοσης από τον ένα τομέα στον άλλο που επηρεάζουν τις προβλέψεις. Όλες οι προβλέψεις για τις χώρες αυτές είναι ε, ε, βασικές προβλέψεις που συζητάμε με τις ενδιαφερόμενες χώρες και με τα θεσμικά όργανα. Επίσης έχουμε και διαφορετικά σενάρια αλλά το βασικό σενάριο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για την πολιτική μας. Να περάσω στην Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα οι διαφορές μεταξύ των προβλέψεων και των αποτελεσμάτων ήταν μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες χώρες ενδεχομένως ε, ε, έχουν γίνει λάθη εδώ, σε άλλες περιπτώσεις τα πήγαμε καλύτερα για την Ελλάδα. Είναι σαφές ότι για την πρώτη χρονιά, αν κοιτάξουμε το αποτέλεσμα και τα, ε, τις προβλέψεις ήμασταν πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από τον πρώτο χρόνο του ε, προγράμματος. Ε, είχαμε μια εκτενή συζήτηση. Τι εννοείται? Το περιβάλλον στο οποίο κινήθηκε το πρόγραμμα ήταν εντελώ διαφορετικό από ό,τι ήταν στην αρχή. Η οικονομική κατάσταση στην ε, περιοχή του ευρώ, στην ε, ε, οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα δεν μπορεί κανεί να τα προβλέψει και να κάνει σωστέ προβλέψει όπω στην περίπτωση τη Ελλάδα. Έχουμε απόλυτη συνείδηση αυτού και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να περιορίσουμε αυτό στο μέλλον. στην Κύπρο ξέρουμε ότι υπάρχουν αβεβαιότητε. Εδώ έχουμε προβλέψει μια μείωση Τη ανάπτυξη κατά 8%. Ε, τώρα ε, ε, είναι κάτι που, για το, το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε με το συντηρητισμό και την απεσιοδοξία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Η εντολή τώρα, όπω σα είπα, η εντολή προέρχεται από τις χώρες μέλη και από το Eurogroup. Αν, υπάρχει, αν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, διεξάγεται μια συζήτηση, ε, ε, το, το ε, θέμα συζήτησης από την ε, Επιτροπή, από τις χώρες μέλη και κατά τη διάρκεια των αποστολών υπάρχει μόνιμη επαφή μεταξύ των επικεφαλής των αποστολών και της, ε, του επικεφαλής της ε, ομάδας της. Υπάρχει συνεπώς, διεξάγονται πάρα πολλές συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων. Μην, μην μου λέτε λοιπόν ότι ε, δρούμε σε ένα κενό. Από την αρχή υπάρχει απόλυτη κατανόηση του τι είναι το πρόγραμμα και υπάρχει μια διαρκής, ένας διαρκής έλεγχος αυτού και σε τελική ανάλυση το, μνημόνιο συζητιέται με τις χώρες μέλη και εγκρίνεται από το Eurogroup. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία όπου εμπλέκονται όλες οι χώρες μέλη. Δεν είναι κάτι που κάνουμε μόνοι μας χωρίς να έχουμε κάποια ανατροφοδότηση, χωρίς να έχουμε ενδείξεις ή χωρίς να έχουμε ε, οδηγίες από τις χώρες μέλη. Τελευταίο σημείο αφορά το... Όχι, όχι, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Ε, κοιτάξτε, ε, ο, χρο... ο, τρόπος που υπολογίζετε το χρόνο σας ε, θυμίζει λίγο τον τρόπο με τον οποίο κάνετε τις προβλέψεις σας. Δεν φταίω εγώ, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πάρω τη σκητάλη από το Σερβάς και να συμπληρώσω στα λεγόμενά του. Να μιλήσω καταρχάς για τις ε, προβλέψεις. Εκ των υστέρων μπορεί κανείς να υποφεληθεί από την εμπειρία. Ως προς τις ελληνικές προβλέψεις σίγουρα μπορεί κανείς να πει ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά και θα έπρεπε να είχαν γίνει διαφορετικά. Πρέπει να αξιολογούνται οι προβλέψεις λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία τη στιγμή που έγιναν οι προβλέψεις. Βάσει των στοιχείων λοιπόν στην Ελλάδα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2010 ε, προβήκαμε σε προβλέψεις για το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής. Τα στοιχεία ήταν ατελή, ε, ελληματικά. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2010, το έλλειμμα για την προηγούμενη χρονιά υποτίθεται ότι θα ήταν 12-12,5%. Ε, μπορεί να ασφάλω εκεί, αλλά εν πάση πτώση είναι σίγουρα πάνω από 10. Μετά από 1,5 χρόνο το στοιχείο αυτό ήταν λοιπές, είχε πάει στο 15,6%. Μεγάλη διαφορά. Ε, ε τεράστιος αντίκτυπος. Δεν είχαμε ακριβή στοιχεία για την ακριβή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και την, το ακριβώς μέγεθος, αν θέλετε, του δημοσίου τομέα. Από εκεί και πέρα, είναι αληθές ότι την άνοιξη του 10 δεν είχαμε γνώση του βάθους των διαρθρωτικών και θεσμικών προβλημάτων που είχαν συσσωρευτεί στη χώρα αυτή. Πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ε, για τις οποίες είχε συμφωνήσει και τις είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Και είχαμε ε, αυτή την κατάσταση το 2012 η οποία υπονόμευσε την εμπιστοσύνη εξού και υπήρξε πολιτική κρίση από πέρα από την έλλειψη ε, από την αδυναμία εφαρμογής των συμπεφωνηθήσεων μεταρρυθμίσεων. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί αθρηστικά ε, ε, εξηγούν την απόκληση στις προβλέψεις και στα αποτελέσματα. Και τέλος, οι αρχές στην πλειονότητα των περιπτώσεων ήταν πολύ πιο αισιόδοξε. Κάθε φορά που πηγαίναμε στην Αθήνα έλεγαν ότι οι δικές μας προβλέψεις είναι εξαιρετικά απεσιόδοξες. Οι προβλέψεις που προβάλαμε εμείς στην αρχή του προγράμματος. Αυτά για αυτό το θέμα. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις για το κατά πόσο υπάρχει ε, φως ε, στο τούνελ κατά πόσο η έξοδος είναι κοντά. Σίγουρα τα στοιχεία για την απασχόληση είναι δίκτες. Δεν μας εκπλήσει. Είναι δυστυχές, αλλά δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι η ανεργία δεν μειώνεται είναι σταθερή, έχει αρχίσει να μειώνεται η ανεργία μόνο στην Ιρλανδία. Οι άλλοι δείκτες όμως, η ανταγωνιστικότητα, ε, η ουσιαστική μείωση του ελλείμματος του κράτους, ε, η ενίσχυση των, ε, των βιβλίων των τραπεζών, το ότι γίνονται πιο δυνατές από λογιστικής πλευράς. Αυτοί είναι δείκτες σημαντικοί και μας κάνουν να υποστηρίζουμε τις προβλέψεις που έχουμε για τα επόμενα χρόνια και για τον αποπληθωρισμό και την ε, μείωση των μισθών. Ε, σε ορισμένες χώρες όντως ισχύει. Υπήρχε αποπληθωρισμός, πέφτουν οι τιμές, σε άλλες όχι τόσο. Στη ζώνη του ευρώ, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, στη ζώνη του ευρώ, αν οι τιμές σε μια χώρα πέφτουν θα πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Και αυτό δεν είναι κακό αυτό αυτό. είναι καλό. Οι καταναλωτές θα έχουν χαμηλότερες τιμές για δεδομένο ονομαστικό μισθό. Και όταν πέφτουν οι τιμές σε σχέση με τον ονομαστικό μισθό, οξύνεται, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας αυτής εναντί των υπολείπων. Ε, άλλο η σχετική αλλαγή τιμών, και αυτό είναι ευχάριστο να συμβαίνει στην Ελλάδα γιατί πρέπει η Ελλάδα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και άλλο αυτό που συμβαίνει στη ζώνη του ευρώ συνολικά όπου δεν υπάρχει αποπληθωρισμός στην ευρωζώνη ως σύνολο. Και ε, ε, τελικά για τις προβλέψεις. Όντως εσφάλαμε. Ε, έχουμε εσφάλει στις προβλέψεις για την Ελλάδα και εξήγησα τους λόγους. Όμως στην Ιρλανδία στις προβλέψεις μας πέσαμε μέσα. Δεν πέσαμε έξω έχουμε τον ιδιωτικό τομέα στην Ιρλανδία και συζητούσαμε με τις Ιρλανδικές αρχές το κατά πόσο η εφαρμογή του μνημονίου στην Ιρλανδία και του προγράμματος θα οδηγήσει τη χώρα σε, μια σε ένα βιώσιμο χρέος και δεν θα χρεοκοπήσει η χώρα αυτή και αυτό επαληθεύτηκε. Οι προβλέψεις λοιπόν για τον ιδιωτικό τομέα στην Ιρλανδία είναι πολύ καλύτερες τώρα. Ε, είναι όντως δύσκολα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει το επιχείρημα ότι η Τρόικα δεν έχει καλές ε, προβλέψεις και ότι δεν κάνει τη δουλειά της σωστά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ξέρετε, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο άκουσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχουμε το λάθος πληθωρισμό. Ενώ τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας λέει ότι σε ορισμένε χώρες έχουμε το σωστό είδος αποπληθωρισμού. Λες και μιλάμε για καλή και κακή χολυστερίνη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στι στις τελευταίες τρεις ερωτήσεις. Λάγγεν, Θέο και Ποδηματά. Παρακαλώ. Um, και θα υπάρξει διερμηνία για τις ερωτήσεις, αλλά ίσως δεν θα υπάρξει και για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από τις πολλές ερωτήσεις θα είμαι σύντομο που έχουν γίνει ήδη. Έχετε μία εντολή από τους Υπουργούς Οικονομικών, από την Κομισιόν, γιατί αρνήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι σήμερα μαζί σας. Μήπως αυτό οφείλεται σε διαφορετική εκτίμηση της κατάστασης. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, αν δείτε το παρελθόν, μιλήσατε για τις προβλέψεις σας, δεν ε, είναι εύκολο να κάνει κανένας προβλέψεις παρά μόνο με σωστά στοιχεία. Τι θα κάνατε διαφορετικό σήμερα με την εμπειρία των τελευταίων τριών ετών. Πού θα κάνατε κάποια διαφορά σε σχέση παραγωγός χάρη με τις προβλέψεις σας για την κίνηση των μισθών και των τιμών. Και το τρίτο ερώτημα, πώς λειτουργήσε η, η συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε κάθε χώρα που, του προγράμματος. Ο Διόγκο Φέου. Ευχαριστώ Σέρον. Εγώ θέλω να τονίσω καταρχήν ότι Συμφωνώ ότι οι χώρες που δεν είχαν τους δημόσιους λογαριασμούς σε καλή κατάσταση έπρεπε να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Αλλά δεν καταλαβαίνω όταν λένε ορισμένοι σήμερα κάποιοι βουλευτές από κόμματα που ήταν στην κυβέρνηση και αυτό συνέβη στην Πορτογαλία που ξέραν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα και ήταν απαραίτητο το πρόγραμμα ε, προσαρμογής τώρα να μιλάνε σαν να μην ήταν καθόλου απαραίτητο. Μίλαμε τώρα για την ανάγκη βοήθεια σε χώρες οι οποίες είναι σε κρίση. Το κύριο πρόβλημα των προγραμμάτων αυτών είχε να κάνει με το κοινωνικό επίπεδο. Είναι τεράστιος ο αριθμός, είναι ανησυχητικός ο αριθμός των ανέργων στις χώρες αυτές της κρίσης. Και θα ήθελα να ξέρω σε σχέση με αυτούς τους αριθμούς, αν η Κομισιόν και η Κεντρική Τράπεζα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα προγράμματα αυτά ήταν σωστά σχεδιασμένα ή αν παραδέχονται ότι υπήρχαν σφάλματα σε αυτά τα προγράμματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Δεύτερον, είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις θέλαν να υπάρχει μεγαλύτερη ευκαμψία στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Ποιοι και ότι οι διεθνείς φορείς Ορισμένοι διεθνεί φορεί τόνισαν ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευκαμπιστοποίηση των προγραμμάτων. Γιατί δεν δεχτήκατε εσεί όμω μια τέτοια ευελιξία. Και έχουμε εξάλλου χώρε που είναι σε τελείω διαφορετικέ συνθήκε. Υπήρχε πρόγραμμα, πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ε, Ιρλανδία και στην ε, Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα και την Πορτογαλία υπήρχε πρόβλημα παραγωγικότητα. Γιατί χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρότυπο για να μπορέσουν να γίνουν οι προσαρμογές στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ Σάρων. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και πάρα πολύ συγκεκριμένη. Το ερώτημά μου είναι προς τον κύριο Ντερούζ. Κύριε Ντερούζ, όπως ξέρουμε, αυτή η συζήτηση είναι πραγματικά επίκαιρη, γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινάει ακόμα μία επισκόπηση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει. Όπως είπατε, η Ελλάδα θα επιτύχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ήδη στο τελευταίο μέσα στο 2013, πιο νωρίς από ό,τι προβλεπόταν και ξέρουμε ότι η Κομισιόν έχει διαμφισβητήσει το κατά πόσο είναι βιώσιμο αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα και γι' αυτό λέτε ότι θα πρέπει να το επανεξετάσετε, η Eurostat θα πρέπει να το επανεξετάσει και να το εκτιμήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Το ερώτημά μου είναι, είναι πώς θα γίνει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα βιώσιμο. Πιστεύετε ότι χρειάζονται περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα, γιατί αυτό είναι που είναι υποσυζήτηση στην Ελλάδα. Με περαιτέρω μείωση των πόρων που πηγαίνουν στην πραγματική οικονομία, μπορούν αυτά να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και πώς και πότε θα έρθει η οικονομική ανάκαμψη. Και τέλος, ένα ερώτημα που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι. Εσείς λαμβάνετε υπόψη το κοινωνικό και το πολιτικό κόστος, τη διάσταση της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας που είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιτυχή εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε στις απαντήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς, οι οποίοι μας έδωσαν ένα τέταρτο πρόσθετο και πρέπει να φύγουν τώρα.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 γνωρίζετε θα υπάρξει ένα μικρό πλεόνασμα τώρα του, του πρωτογενούς. Όπως ξέρετε ο στόχος είναι 4,5 για να είναι βιώσιμο το χρέος. Αρκετά έχουν ε, γίνει. Έχουμε φτάσει στο 13-14% αλλά πολλά μέλουν να γίνουν ακόμα. Πιστεύω ότι πολλά θα προκύψουν από την ίσπραξη φόρων, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κτλ. Τελευταίο σημείο αφορά τον κοινωνικό κλάδο. Ένα σημαντικό σημείο κυρία Πρόεδρε. Στα πλαίσια του προγράμματος δίνεται μεγάλη προσοχή σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα. Έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι θα πρέπει να γίνει καταμερισμός του άχθους. Ξέρουμε ότι όταν υπάρχει μία αντίληψη, αδικίας είναι κακό για την οικονομία, και έχει υπονομεύει την πολιτική στήριξη. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν ο κοινωνικός τομέας. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι σημαντικό στοιχείο όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα της οικονομίας αλλά και για την πολιτική στήριξη της οικονομίας. Αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να τονίσουμε σε όλες τις χώρες αυτές υπάρχουν μέτρα που ελαφρύνουν το, το άχθος. Ε, έγιναν ε, περικοπές αλλά οι ομάδε αυτέ θα τύχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Υπάρχει, καταβάλλονται προσπάθειες για το κοινωνικό δίκτυο. Υπάρχει, καταβάλλονται ιδιαίτερε προσπάθειες στην Ελλάδα και θα γίνουν περαιτέρω προσπάθειες με την Παγκόσμια Τράπεζα. Υπάρχουν μέτρα για τη βελτίωση των κοινωνικών παροχών. Για παράδειγμα, όλα ε, ο τομέα ε, τη υγειονομική ε, περιθαλψη έχει στόχο την καλύτερη ε, χρηματοδότηση και τη μεγαλύτερη πρόσβαση. Επίσης και αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα που έχει συνυπολογιστεί στο πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι σύμφωνα με την Ιρλανδική κυβέρνηση τα προγράμματα κοινωνικής αρρωγής βοήθησαν ιδιαίτερα ε, στον τομέα των κοινωνικών παροχών αυτό ε, οι Ιρλανδοί θεωρούν ότι δίκως αυτό το πρόγραμμα θα είχαν πληγεί κοινωνικές υπηρεσίες. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά απλά και μόνο παρέθεσα ορισμένα παραδείγματα για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο μας απασχόλησε ο κοινωνικός τομέας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ μπορώ να είμαι πιο σύντομος γιατί ο προλαλής σας αναφέρθηκε στα θέματα πάρα πολύ εκτενώς. Θα ήθελα να προσθέσω Να πω κάτι για την κοινωνική διάσταση και το, να απαντήσω το ερώτημα τι θα κάναμε διαφορετικά. Ίσως από την αρχή και σκέφτομαι τώρα για την Ελλάδα θα, είχαμε, θα έπρεπε να είχαμε θέσει μεγαλύτερη πίεση στην ε, μεταρρύθμιση της αγοράς προϊόντων. Μας εξέπληξε πόσο μεγάλη ε, αντίσταση υπήρξε και πόσο ισχυρά ήταν κάποια επενδεδημένα συμφέροντα. Αυτά τα συστήματα λοιπόν ε, για την αποδυνάμωση των μεταρρυθμίσεων και την αντίσταση των μεταρρυθμίσεων είναι αυτοί οι οποίοι είναι βολεμένοι και οι οποίοι προστατεύουν τον εαυτό τους, είναι τα άτομα υψηλού εισοδήματος, είναι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίας κτλ. Το να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν μια ε, ακύρωση των προνομίων που επιτρέπουν σε ορισμένους να κρατάνε υψηλά τις αμοιβέ τους και υψηλά, υψηλά τις τιμές σε βάρος των καταναλωτών. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και το είχαμε στην αρχή στο πρόγραμμα για την Ελλάδα, αλλά μετανιώσαμε μετά. Δεν υπήρξαν πολλές προτάσεις από την πλευρά της κυβερνήσεως και κατά τη διάρκεια της, ε, του προγράμματος κάναμε προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά και βέβαια βοήθησαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη. Τα θέματα της ε, διοίκησης είναι άλλες περιπτώσεις όπου η φοροδιαφυγή πράγματι και η φοροαποφυγή υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν την δικαιοσύνη της ε, φορολογίας και να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ. Και ο κύριος ε, Δερός έχει δώσει πολύ καλά παραδείγματα των προσπαθειών μας όταν συζητούμε με την κυβέρνηση και λέμε ότι πράγματι ανησυχούμε για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν και είναι οι πιο τροωτοί και έχουμε ένα κοινό στόχο όταν συζητούμε με τις κυβερνήσεις για να ξεπεράσουμε τη κρίση, να τελειώσει η κρίση το ταχύτερο δυνατό και να δημιουργήσουμε τα θεμέλια για, για μεγαλύτερη η ανάπτυξη και να κάνουμε πιο αθεκτικές οικονομίες μας <clears throat> για να αντιμετωπίσουν μελλοντικού κλειδονισμούς γιατί οι ακαμψίες τους των χωρών αυτών αυξάνουν το κοινωνικό κόστος της κρίσης και της ανεργίας και δεν θέλουμε να έχουμε το ίδιο πρόβλημα όταν έχουμε την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση η οποία θα επανέλθει ίσως ή θα επανέλθουν κλειδονισμοί τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο ανθεκτικοί ώστε οι χώρες αυτές να μπορέσουν να αντέξουν περαιτέρω κλειδονισμούς χωρίς τόσο μεγάλο κοινωνικό κόστος. Αυτό είναι ο κοινό μας στόχος της Τρόικα και πιστεύουμε ότι αυτό το συμμερίζονται και οι αρχές των χωρών αυτών και οι υπουργοί τη Ευρωομάδα και οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ μα. Θα μπορούσαμε να περάσουμε όλο το απόγευμα με κάθε μέλο του πάνελ. Συγγνώμη που σα έχουμε πιέσει χρονικά. Έχουμε όλοι του ίδιου στόχου να τελειώσει η κρίση και να επανέλθουμε στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Είναι σαφέ όμω ότι <clears throat> η συμμετοχή των λαών και των κοινοβουλίων ε, απαιτεί καλύτερη πληροφόρηση και όχι μονάχα εκ των υστέρων να μαθαίνουμε τι έχει γίνει. Θα συζητήσουμε και πάλι για τα θέματα αυτά στο μέλλον.